Eh, Γεια σας, καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας, τη σημερινή. Έχουμε ένα απόγευμα πολύ ενδιαφέρον μπροστά μας με, με ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πρώτα απ' όλα θα συζητήσουμε σε υψηλό επίπεδο διάφορα θέματα που αφορούν το mainstreaming που θα πρέπει να εφαρμόσουμε εδώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν τέτοιε αιτήσει αλλαγή, μπορούμε να δεχτούμε την ημερησία διάταξη. Περνάω στι ε, ανακοινώσει τη Προέδρου και μέσα στι ανακοινώσει αυτέ θέλω να σα παρακαλέσω να τηρήσετε στρατιωτική πειθαρχία. Γιατί έχουμε πολλά θέματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε σήμερα. Προετοιμάζοντας τις ε, Ολομέλειες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, ιδίω στο Στρασβούργο, και θα ήθελα να το καταγράψει αυτό ότι είναι απαραίτητη η παρουσία σας στις Ολομέλειες αυτές και στην ατζέντα σας. Πάω στο σημείο 3 τώρα ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη που είναι υπεύθυνα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να καλωσορίσω και την κυρία Κόχ Μεϊρίν η οποία είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιπλέον είναι η πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μας να συζητήσουμε και το θέμα αυτό, όπως είχαν ζητήσει και τα μέλη μας τα οποία ασχολούνται με τα θέματα της ισότητας των φύλων. Είχαμε ήδη, ήδη το Μάρτιο μία συνάντηση και εκεί είχε διατυπωθεί και η αίτηση να έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους στόχους που επιζητεί η ομάδα υψηλοπιπέδου για την ισότητα των φύλων και τις ε, και της ε, ε, ισότητας ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα, όχι και γυναικών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα <clears throat> από την πλευρά της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κοχμέριν που έχετε έρθει στη συνεδρίασή μας και ασμένως σας δίδω τον λόγο ώστε να μπορέσετε να μας πληροφορήσετε για το έργο της ομάδας σας υψηλού επίπεδου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Αγαπητές συνάδελφοι, νομίζω ότι δεν υπάρχουν άρενες βουλευτές εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι μπορούμε να προωθήσουμε τη συνεργασία μας μεταξύ της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ισότητα των φύλων και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών, όπως τόνισε και η πρόεδρος, η οποία είναι και αυτή μέλος σε αυτή την Επιτροπή Υψηλοπιπέδου, σε αυτήν την ομάδα Υψηλοπιπέδου, γνωρίζει επομένως ότι στους επόμενους, μάλλον στους πρώτους 12 ή 15 μήνες κατά τους οποίους εργάστηκε η ομάδα μας, έχουμε ήδη προχωρήσει σημαντικά και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε και πιο εντατικές πρωτοβουλίες. Καταρχήν δύο λόγια για το τι είναι η ομάδα αυτή υψηλοπιπέδου, τι κάνει, ποιοι είναι οι στόχοι τη, και γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο να υπάρχει καλή συνεργασία με αυτή την ομάδα, της Επιτροπής σας με αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι στη συντριπτική μας πλειοψηφία τα μέλη της ομάδας μας επιζητούν τους ίδιους στόχους, δηλαδή να υπάρξει απόλυτη ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών, να υπάρξει αναγνώριση και σεβασμός της διαφοράς ε, σε ό,τι αφορά τη θρησκεία ή την ε, σεξουαλική προτίμηση σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα όμως της Επιτροπής μας, εμείς περιοριζόμαστε στα θέματα της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή με τις δεδομένες τομές οι οποίες υπάρχουν στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά έχουμε σημαντικούς στόχους, διότι το Κοινοβούλιο μας έχει διατυπώσει πολλές φορές συγκεκριμένους στόχους, παραγωγός χάρη τα θέματα της συμβατότητας επαγγελματικής και οικογενειακή ζωής ή οι δυνατότητε, οι πιο ηλικιωμένε γυναίκες να παραμένουν στον χώρο της εργασία. Όλες αυτές οι δυνατότητες λοιπόν, που έχουν να κάνουν με την ε, ισότητα των φίλων και των ευκαιριών στην κοινωνία είναι στόχοι που πρέπει να τους επιτύχουμε και για μένα ένα σημαντικό σημείο της αξιοπιστίας της δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αυτοί οι στόχοι να επιτυγχάνονται και στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί τότε μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οποίο ζητούμε για τους άλλους το έχουμε ήδη εδραιώσει και επιτύχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επομένω έχουμε μια σαφή και απτή αντιμετώπιση. Επομένω, η ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου έχει να κάνει με την εφαρμογή αυτών των στόχων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλει να δώσει σάρκα και οστά σε αυτέ τι διακεκηρυγμένε αρχέ και να μπορέσει να τι εφαρμόσει στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κάνουμε αυτό με τη χρήση διαφόρων εργαλείων και μέσων. Έχουμε καταρχήν ένα σχέδιο δράσης. Κάθε χρόνο καταρτήσουμε ένα σχέδιο δράσης με ενημέρωση και επικαιροποίηση των στόχων μας και έχουμε ήδη εγκρίνει ένα πολιετές σχέδιο δράσης που καλύπτει το χρονικό διάστημα 2009 έως 2013 και έχει χαράξει τις κύριες κατευθυντήρες γραμμές μέσα στις οποίες θα επακολουθήσουν τα ετήσια σχέδια. Έχουμε επίσης δημιουργήσει και ένα δίκτυο για την συμπερίληψη όλων των θεμάτων που άπτονται της διάστασης των φύλων, που συνδέει όλες τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και επιτροπές με, την, με το συντονισμό της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Εμείς <clears throat> υποστηρίζουμε λοιπόν το να μπορέσουν να υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα ε, στα πλαίσια αυτά, στις επιτροπές και αντιπροσωπείες και επίσης το να υπάρχει αντικατοπτρισμός της ισότητας των ευκαιριών και των φύλων και στη γραμματεία των επιτροπών. Επίσης να εξασφαλίσουμε μία ουδέτερη σε σχέση με τη διάσταση των φύλων γλώσσα σε όλα τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα βέβαια. Ξέρετε ότι σε γλωσσικό επίπεδο σε κάθε γλώσσα είναι διαφορετικά τα θέματα. Στα σουηδικά ξέρω ότι το θέμα αυτό δεν <clears throat> είναι πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει μια τέτοια διάκριση μεταξύ των φύλων σε γλωσσικό επίπεδο αλλά σε πολλές άλλες γλώσσες τα πράγματα είναι διαφορετικά γιατί επικρατεί πάντα η το, το αρσενικό άρθρο ή το αρσενικό κατά κάποιο τρόπο γένος στην, ε, στην διατύπωση των ε, διαφόρων εγγράφων. Έχουμε επίσης μια σειρά από τακτές επαφές με άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι κάτι το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει πάντα και κατ' επανάληψη ότι εμείς θέλουμε να είμαστε το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα αποτελεί και παράδειγμα προς για τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως είναι σημαντικό για να το επιτύχουμε αυτό να έχουμε μια διοίκηση η οποία αντικατοπτρίζει την ισότητα ευκαιριών μεταξύ των φύλων και την πολυμορφία, το σεβασμό της πολυμορφίας και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις στα άλλα ε, θεσμικά όργανα. Η ομάδα εργασία λοιπόν υπάρχει από το 2004 για την ισότητα των φύλων. Όταν δημιουργήθηκε σαν ε, απάντηση κατά κάποιο τρόπο σε μια έκθεση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και στα ετήσια σχέδια δραστηριότητος τα οποία καταρτίζουμε είναι προφανές ότι εμείς ανταλλάσσουμε πάντα απόψει και θέλουμε να έχουμε και τη συμβολή τη Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών, η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά. Η σύνδεση τώρα τη ομάδα μα, υψηλό επίπεδο, εγώ έχω την τιμή να είμαι πρόεδρο αυτή τη ομάδα. παραδοσιακά πρέπει να προεδρεύει αυτή τη ε, ομάδα ένα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι με τον τρόπο αυτό εκπροσωπούμε και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε τη σύνδεση με το Προεδρείο. Η κυρία Αντζελίλη είναι αντιπρόεδρος της ε, ομάδας υψηλού και έχουμε τώρα σαν μέλη την κυρία Ροτ Μπέρεντ, την κυρία Σβένσον επίσης, η οποία έχει διπλή εκπροσώπηση. Επίσης ο κύριος Καρλ Λένε είναι παρόν και ως πρόεδρος επιτροπής, αλλά σίγουρα οι πρόεδροι των Επιτροπών εκπροσωπούνται και από την κυρία Μπριτ Σφένσον, η οποία νομίζω ότι ω πρόεδρο τη Επιτροπή ε, Γυναικών μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ο κ. Παϊνονοεύο επίση ω πρόεδρο εκπροσωπεί την ε, συνέλευση των ε, πρόεδρων των Αντιπρόεδρων. Η κυρία Έντεμπερκ επίση εκπροσωπεί τους ε, Κοσμήτορες, νομίζω ότι ήταν μέλος της Επιτροπής σας. Η κυρία Λούλινγκ επίση είναι μέλος. Ο Πάουλ Σμιτ ήταν ε, μέλος αυτής της Επιτροπής. Βέβαια έχει επιστρέψει ως πρόεδρος της ε, Ουγγαρίας. Και κάνουμε προσπάθειες για να μπορούμε να έχουμε και ένα δεύτερο άντρα στην Επιτροπή μας, ώστε να μπορούμε να συζητούμε όλα αυτά τα θέματα που άπτονται τις ισότητα των μήλων, των φίλων, συγγνώμη. Αυτή είναι λοιπόν μια σύντομη επισκόπηση της σύνθεσης και της δραστηριότητας της ομάδας υψηλού επίπεδου και είμαι έτοιμη να απαντήσω στα ενδεχόμενα ερωτήματα τα οποία έχετε και να δώσω συνέχεια τις προτάσεις και τις συστάσεις τις οποίες θέλετε να διατυπώσετε. Έχουμε τονίσει λοιπόν ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ενσωμάτωση τη ε, ισότητα του φύλου στι πολιτικέ πρωτοβουλίε και στι δραστηριότητε των επιτροπών, το λεγόμενο gender mainstreaming. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει και μια ομάδα εργασίας η οποία καθαρίζει, καθορίζει τις κατευθυντήρες γραμμές για μια ουδέτερη ως προς τα φύλλα γλώσσα, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται και σε εξωτερικό αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο μέσα στην ε, επικοινωνία, μέσα στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρακολουθούμε ακριβώς και ελέγχουμε την, τις διατυπώσεις που χρησιμοποιούνται. Επίσης, στα πλαίσια των επαφών με τα άλλα θεσμικά όργανα έχουμε τακτικές επαφές και με την Κομισιόν, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους ε, φορείς. Και επίσης πολλές φορές προσκαλούμε τους εισηγητές και άλλων θεσμικών οργάνων για τα θέματα αυτά στην ομάδα εργασία μας. Πέντε στόχους έχουμε προς το παρόν στο σχέδιο στο πρόγραμμα εργασία μας, καταρχήν ισότητα ανδρών και γυναικών, Δεύτερον, ίσες ευκαιρίες για τα άτομα τα οποία έχουν αναπηρίε ή ειδικέ ανάγκες. Να αρθούν οι φραγμοί για την πρόσληψη. Να υπάρξει ενίσχυση των ηγετικών θέσεων που πρέπει να είναι πιο ανοιχτές στην πολυμορφία και επίσης δημιουργία ενός πιο περιεκτικού και ολοκληρωμένου περιβάλλοντος εργασίας. Για κάθε στόχο έχουμε συγκεκριμένα εγχειρήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, παραδείγματος χάρη για το πόσες γυναίκες θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε συγκεκριμένο διοικητικό σκαλί της ιεραρχίας. Πρέπει να παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε τώρα ότι αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε επίπεδο πραγματικότητας. Επίσης το ίδιο πράγμα κάνουμε και για τα άτομα τα οποία έχουν αναπηρίες ή άτομα τα οποία έχουν συγκεκριμένες θρησκευτικέ πεπιθήσεις. Και επίσης να εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα τα οποία έχουν ελαφρές αναπηρίες να μην υφίστανται δυσκολίες. Σε ό,τι αφορά τα ανώτατα κλιμάκια, το λεγόμενο senior management level, έχουμε τέσσερις γυναίκες από τα 11 άτομα τα οποία είναι γενικοί διευθυντέ. Αυτό είναι 36%. Δεν είναι άσχημο αριθμό, δεν είμαστε ακόμα στο 50%, αλλά είναι <clears throat> πολύ περισσότερο από ότι ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί που ήταν 20% και τώρα μπορούμε να είμαστε και πιο φιλόδοξοι στην στοχοθεσία μας. 32% γυναίκες στο αμέσως πιο κάτω επίπεδο, που είναι οι διευθυντέ, εκεί ο στόχο ήταν 35%. Δεν το πετύχαμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι πολλέ φορέ στο ενδιάμεσο επίπεδο διοίκηση μόνο 22% των επικεφαλή μονάδων είναι γυναίκε. Και οι αρχηγοί μονάδων είναι αυτοί από τους οποίους προέρχονται πολλές φορές τα ανώτερα κλιμάκια. Επομένως θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στον τομέα αυτό. Έχουμε λοιπόν τους στόχους τους οποίους θέτουμε σε επίπεδο ετήσιο και είχαμε και την πρωτοβουλία την οποία διατύπωσε καταρχήν η κυρία Σφένσεν να υπάρξει και συμπερίληψη της λέξεως ποσοστώσεις. Και αυτό νομίζω ότι έχει θεωρηθεί και από το Προεδρείο και από την Γερική Γραμματεία του Κοινοβουλίου σαν μια οδός η οποία μπορεί να επιταχύνει την οδό προς την ε, ισότητα. Γιατί υπήρχαν στο παρελθόν πολλές περιπτώσεις που δεν υπήρχε ούτε μία γυναίκα μεταξύ των υποψηφίων. Κάτι κατά την απόψή μου δεν είναι καθόλου σωστό. Ελπίζουμε λοιπόν ότι τις επόμενες εβδομάδες στις 16 ε, Νοεμβρίου να έχουμε και το σχέδιο εργασίας για το 2011, το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεχομένω επιχειροποίησεις και αλλαγές στο σχέδιο δράσης μας. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι σας δίνουν μια πρώτη ε, επισκόπηση, μια πρώτη οπτική γωνία για το τι κάνει η ομάδα υψηλοπιπέδου για την ισότητα του φύλου και είμαι έτοιμη να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Stort tack för den här informationen. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάνει η ομάδα υψηλού επίπεδου και εξ ονόματος της Επιτροπής μας πρέπει να ομολογήσω ότι με μεγάλη μας χαρά θα συνεργαστούμε μαζί σας για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ισότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ενημέρωση που μας κάνανε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την ε, συζήτηση. Όπως είπε και η κυρία Κόχμεριν, υπάρχει ένα πρόγραμμα του 2009-2013 και θα πρέπει να συζητήσουμε τώρα τι θα κάνουμε για το 2011. Πρόκειται για ένα κείμενο, για ένα πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε ε, την κατάσταση. Έχετε το λόγο. Η κυρία Λίχθενμπερκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και για την καλή οργάνωση αυτής της ε, ε, συνάντησης. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τακτές επαφές με την ομάδα αυτή υψηλού επίπεδου. Μας ενδιαφέρει πράγματι για πρώτη φορά να εξασφαλίσουμε μια ενισχυμένη συνεργασία για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις γυναίκες και είναι ένα εγκάρσιο θέμα και πιστεύω ότι όλοι οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι ακριβώς λαμβάνει η χώρα και επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διεκδικήσει στα ψηφίσματά του να μπορεί να έχει μια δυνατότητα εφαρμογής. Βέβαια, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση η οποία μπορεί να καλύψει τα θέματα αυτά. Δεν υπάρχει. Πολλές φορές έχουμε απλώς μία διαδικασία. Για τον τομέα αυτό δεν υπάρχει αρκετή συνεργασία και αναφέρομαι στο θέμα των ε, διαζυγίων. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά και στα κράτη-μέλη του σε εθνικό επίπεδο να μας, να μας ε, να κατανοήσουν ότι εδώ δεν είναι ένα θέμα το οποίο οφείλεται σε έλλειψη ρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ακόμα μια αντίδραση, υπάρχει μια ακόμα και αντιδραστική στάση ορισμένων, θα το πω αυτό με κάπως πολεμικό τρόπο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι δεν θέλουν τα θέματα διαζυγίων να βρεθούν σε ένα ευρύτερο, σε ένα ευρύτερο χώρο όπως ο Ευρωπαϊκός στα θέματα των διαζυγίων, τα οποία θέλουν ζηλότυπα να διατηρήσουν σε εθνικό επίπεδο. Είναι δύσκολο να παντρευτεί λοιπόν κανείς και Μαλτέζου αν τα ξέρει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι κι είναι και λίγοι Μαλτέζοι. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και καλύτερη επικοινωνία για τα θέματα αυτά. Η... Θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να θέτουμε ερωτήματα στους εκπροσώπους του Συμβουλίου από τις, από τις χώρες μας γιατί πάντα δεν υπάρχει η προστασία για το ασθενέστερο τμήμα του ζευγαριού που είναι συνήθως οι γυναίκες γιατί δεν υπάρχει λοιπόν αυτή <clears throat> η προστασία και επομένως θα πρέπει να πάρουμε εμείς μια πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε και προς τον έξω κόσμο και να διαδηλώσουμε ότι έχουμε περισσότερες ε, φιλοδοξίες. Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα με τις αναπηρίες όπου θα πρέπει να επιληθεί και η Επιτροπή Μεταφορών, αλλά δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω. Έρχομαι ήδη από ένα ταξίδι αντιπροσωπείας στην Κίνα που κάναμε πρόσφατα και νομίζω και εκεί θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι αντιπροσωπείες όταν μεταβαίνουν στο εξωτερικό για επαφές με τους ομολόγους τους θα πρέπει να τονίζουν πιο έντονα τις ευρωπαϊκές αξίες από τις οποίες εμφορούμεθα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ιδίως σε περιπτώσει όπως τα, για τα θέματα των γυναικών οι οποίε είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενε στις χώρες αυτές και είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τονίζει στεναρά τι απόψει του και να εξασφαλίζει ότι τη χάνουν συζήτηση. Θα ήταν ίσω αυτό ένα σημείο το οποίο θα μπορούσατε να ενσωματώσετε στο σχέδιο εργασία σα για το επόμενο έτος. Ευχαριστώ. Tack Mrs Lichtenberg för de synpunkterna och... Eh, ευχαριστώ για αυτές τις απόψεις. Η κυρία Τόμσον είναι η επόμενη που θα πάρει το λόγο. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την παρουσίαση και αυτό το πρόγραμμα που προτείνατε. το θέμα είναι αυτό της ισότητας των φύλων και χρηματοδότηση βάση του φύλου δεν λαμβάνουμε στη χρηματοδότηση την ισότητα των φύλων. Θα πρέπει όμως να το καταλάβουμε αυτό τι γίνεται όσον αφορά τον προπολογισμό και τα κονδύλια που πηγαίνουν ισότιμα στα φύλλα. Και δεν υπάρχει σε πολλές χώρες ε, επιτροπή γυναικών στο κοινοβούλιο. Στη χώρα μου τη Δανία δεν έχουμε επιτροπή γυναικών και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να γίνουμε έμπνευση εμείς αν γίνουμε πιο ορατοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάτι που είναι πολύ σύγχρονο και προχωρημένο είναι αυτό που λέτε για πρόθεση ανοιχτού περιβάλλοντος που εντάσσονται όλοι εκεί διότι μπορούμε να έχουμε ποσοστώσει συχνά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση για τις γυναίκες στην έρευνα πράγματος χάρη αλλά φεύγουν οι γυναίκες διότι το περιβάλλον δεν, τις, δεν ευνοεί την ένταξη, υποστηρίζει περισσότερο τους άντρες. Οπότε δεν αρέσει στις γυναίκες να μείνουν εκεί και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το περιβάλλον το οποίο να εντάσσει τους πάντες. Θα ήθελα να ξέρω αν βλέπουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την παρακολουθούμε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε για τη χάρτα των γυναικών τον Μάρτιο. Και υποσχέθηκε ότι και 27 επίτροποι θα κάνουν προσπάθεια να συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου στην, στις διάφορες πολιτικές. Νομίζω ότι πολύ συχνά σε διάφορες επιτροπές και στις συζητήσεις και νέες πρωτοβουλίες λείπει η διάσταση του φύλου και όταν συζητάμε νέες ε, οδηγίες. Σας ευχαριστώ κυρία Τόμψεν. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπόουερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω κι εγώ. Είναι καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν το θέμα της ισότητας των φίλων στο Κοινοβούλιο. Οπότε έχω ένα ερώτημα σχετικά με το θέμα που συζητούμε. Αναφέρθηκε λοιπόν η αυξημένη διευρυμένη συνεργασία. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, όπου συμμετέχει η Επιτροπή Γυναικών, κάθε φορά που συζητείτε, πώς να το πω, δεν συζητείται με τον δέοντα τρόπο. Ίσως έτσι μπορώ να το θέσω. Καμιά φορά οι συζητήσεις παίρνουν παράξενη μορφή και τόνο. Θα ήταν δυνατόν να ασχοληθούμε με το ζήτημα στην ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου καμιά φορά και όταν θα χρειαζόταν. Η διάσταση του φίλου να ε, χρησιμοποιηθεί και να εξεταστεί και σε αυτή την περίπτωση ακόμα η διαβριμένη συνεργασία δεν είναι πολύ ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπάουερ. Η κυρία Ματέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εδώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο όπως και οι άλλες συνάδελφοι γιατί είναι πολύ καλό που υπάρχουν πάντοτε τέτοιες συναντήσεις που μας ναι. επιτρέπουν να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να αναφερθούμε και σε αυτές τις πέντε προτεραιότητες του προγράμματος δράση. Θα ήθελα να ξέρω επίσης η προσοχή την οποία θα πρέπει να αποδώσουμε στην ισότητα αμοιβών ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, κυρίως αναφορά αφορά τις συντάξεις Πού θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το εντάξουμε, γιατί η Κομισιόν το έχει συζητήσει μέσα στα πλαίσια των, της γενικότερης πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι τα θέματα αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών μεν, αλλά η πράσινη βίβλος ε, αφήνει κάποια περιθώρια για κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Επομένως, η ερώτηση που θέτω είναι σε ποια από αυτές τις πέντε κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαμε ε, να συζητήσουμε για, τις, ε, την διαφορά ε, ανάμεσα στις συντάξεις ανδρών και γυναικών. Eh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ματέρα. Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που ακούσαμε. οι συνάδελφοι εκφράστηκαν ιδιαίτερα ευνοϊκά σε σχέση με τις πέντε προτεραιότητες τις οποίες αναφέρατε. Τώρα, ε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να απαντήσετε στα θέματα αυτά. Κυρία Κόχ Μερίνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για τα ερωτήματα και για τις παρατηρήσεις σας. Ίσως έχω ένα μικρό πρόβλημα να απαντήσω όλα αυτά τα οποία θέσατε. Πολλά από αυτά τα οποία αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά δεν εντάσσονται καθόλου στην εντολή της ομάδας εργασίας μας. Εμείς απλώς ασχολούμεθα με το θέμα της γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προφανώς και αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα, γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε τη δίκηση του Κοινοβουλίου σαν χωριστή από τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά θέματα, παραδείγματο χάρη, όπως το δικαίωμα διαζυγίου. Αυτά μπορεί να αφορούν κάποια άτομα, ίσως στην ε, γραμματεία του Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω ότι ίσως είναι μικρό το ποσοστό το, το ποσοστό των ατόμων που Φύγονται από αυτό. Ακόμα και αν είναι πιο μεγάλο το ποσοστό των μεικτών γάμων στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι στα εθνικά κράτη. Αλλά δεν είναι θέμα της ομάδας εργασίας υψηλού επίπεδου να επιληφθεί των θεμάτων αυτών. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βέβαια, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται περισσότερο στα ε, αγροτεμάχια τη Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε την καλή συνεργασία μεταξύ της ε, δικής μας ομάδας υψηλού επίπεδου και της δικής σας επιτροπής. Εγώ φυσικά <clears throat> καταγράφω αυτό το οποίο αναφέρατε, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα συμπερίπτωσης θεμάτων ειδικών με την προβληματική της ισότητας των γυναικών και στις αντιπροσωπίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς μπορείτε φυσικά να το υποστηρίξετε και ως συντονίστρια του δικτύου που περιλαμβάνει αντιπροσωπείες <clears throat> και επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε προφανώς να το υποστηρίξετε. υπάρχει λοιπόν περισσότερη προβληματική για τα γυναικεία θέματα. Επομένως νομίζω ότι και πάλι η πρωτοβουλία δεν πρέπει να έρθει από τη δική μας πλευρά, αλλά από τη δική σας πλευρά. Τώρα, για τις σκανδιναβικέ χώρες νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη και ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Μου κάνει, θα, μου κάνει, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που λέτε ότι δεν υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές για τα θέματα των γυναικών. Το θέμα του gender budgeting, του προϋπολογισμού επί τη βάση των φύλων. Επίσης είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί περιλαμβάνει <clears throat> και την απαραίτητη κατανομή αρμοδιοτήτων και την ισορροπία δυνάμεων. Επομένως το gender budgeting είναι μια σημαντική πτυχή της όλης προβληματικής. Κάτι ακόμα το οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ε, μέτρων τα οποία ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνονται περισσότερες δυνατότητες ακριβώς για αυτό το gender budgeting να έχουμε παραγωγή χάρη μεγαλύτερες δυνατότητες για την ε, εργασία των γυναικών που έχουν οικογένειες οι οποίες είναι πολλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι το 80% των ε, εργαζομένων γυναικών. Επίσης, για το θέμα της άδεια ανεφαποδεχών, του sabbatical. Εδώ δεν έχουμε ακόμα αρκετά στοιχεία για το πώς, οι άνδρες και πόσες γυναίκες παίρνουν αυτή την άδεια για να ασχοληθούν με την οικογένειά τους. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το εξασφαλίσουμε, να το ελέγξουμε και να δούμε ότι να βρούμε τρόπου, η συμφιλίωση οικογενειακή και επαγγελματική ζωή να μην αφορά σχεδόν αποκλειστικά μοναχά τι γυναίκε, αλλά να μπορεί να ενδιαφέρει και του άνδρες. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στο, στο σχέδιο δράση μα. Ένα άλλο σημείο είναι το να υπάρχει ειδική κατάρτιση των γυναικών οι οποίε διεκδικούν μια προαγωγή, θέλουν να ανέβουν στο υψηλ, σε υψηλότερα ε, κλιμάκια της ιεραρχίας και είναι απαραίτητη να υπάρχει μια ειδική υποστήριξη για τις γυναίκες στις προσπάθειες τους αυτές. Τώρα το αν παρακολουθούμε αυτά τα οποία κάνει η Κομισιόν. Βεβαίως. Εμείς έχουμε επαφές με τον κύριο Σεύκοβιτς, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τον προσκαλέσουμε τον Φεβρουάριο σε μια συνάντησή μας. Επίσης έχουμε επαφές με την κυρία Ρέντινγκ, η οποία είναι σαφώς ότι είναι υπέρμαχος και αγωνίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και μπορούμε ίσως να σκεφτούμε και λίγο περισσότερο για τα θέματα των ποσοστώσεων, ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η τελευταία συνάντηση που είχαμε την κυρία Ρέντινγκ. Και ο κύριος Μπούζεκ θεώρησε ότι είναι καλές οι ποσοστώσεις από αυτή την άποψη. Πιστεύω λοιπόν ότι και στην Επιτροπή σας υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία θέλουν να επιτύχουν ακριβώς αυτούς τους στόχους. Κυρία Μπάουερ, αυτά που είπατε για την πιο έντονη συνεργασία μεταξύ μας. Αυτό είναι φυσικά ένα από τα κεντρικά θέματα της δραστηριότητές μας και ισχύουν τα ίδια τα οποία είπαμε την κυρία Λίχτεμπεργκ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με τη γενική πολιτική εργασία και λιγότερο με αυτά που τα οποία κάνουμε μέσα στην διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον είναι να πάρουμε εμεί τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ορισμένες ρυθμίσεις διαθεσμικού χαρακτήρα οι οποίες αντανακλούν αυτές τις ε, ε, κατευθύνσεις που χαράζονται. Κυρία Ματέρα και εσείς αναφερθήκατε στο θέμα της ανισότητος αποδοχών γυναικών και ανδρών και τη μειονεκτική θέση που, στην οποία βρίσκονται πολλές φορές οι γυναίκες. Για μας είναι ένα τελείως έμεσο θέμα γιατί στην ε, δίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει απόλυτη μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν τέτοια ανισότητα αποδοχών, αλλά θέλουμε ακριβώς να εξασφαλίσουμε με την ειδική κατάρτιση των γυναικών για την ε, προαγωγή τους και για την ιεραρχική τους άνοδο, όταν επίσης υπάρχουν διαδικασίες επιλογής υποψηφίων, γνωρίζουμε ότι ορισμένες Θέσει ορισμένε τοποθετήσει, όπω παραδείγματο χάρη να είναι κανεί στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο, στη Washington, και που είναι κάτι το οποίο προωθεί και την ιεραρχική ανέλυξη, βλέπουμε ότι εκεί έχουμε σχεδόν πάντα μόνο άντρε. Ποτέ δεν έχουμε γυναίκες. Μήπως θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική διατύπωση της προκήρυξης. Μήπως θα πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο να το κάνουμε αυτό. Αλλά δεν έχουμε γυναίκες υποψηφίους σε αυτές τι περιπτώσεις. Επομένως, ίσως θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού τομέα. Γιατί και ο ιδιωτικός τομέας έχει αντίστοιχα προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα λύσει. αν θέλετε, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να μην ήταν αρκετά φιλόδοξο ώστε να προχωρήσει σε πιο ανορθόδοξες μεθόδους για να εξασφαλίσει την ισότητα ανδρών και γυναικών. Και εγώ θα πρέπει να περιλαμβάνουμε στην προκήρυξη των θέσεων αυτών το ότι πρέπει να υπάρχει και ένας επαρκής αριθμός γυναικών υποψηφίων και να μην μπορεί να προχωρεί μια διαδικασία μονάχα με άντρες. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές συνθήκες από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά σίγουρα εμείς έχουμε ε, την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σαν δημόσιος τομέας. Και βλέπετε και στον ιδιωτικό τομέα ότι όταν θέλουν οι εταιρείε να εξασφαλίσουν μια ισότητα ανδρών και γυναικών, θα πρέπει να κάνουν κάποια θετικά μέτρα προ την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και για να κλείσουμε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ξανά ότι αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου ασχολείται με διοικητικά θέματα και η δική μας Επιτροπή ασχολείται επίσης με θέματα πολιτικά. Υπάρχει σχέση μεταξύ των διοικητικών μέτρων και της δουλειάς που κάνουμε στην Επιτροπή, άρα είναι σημαντικό να βλέπουμε συνολικά τα πράγματα, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να τα βελτιώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες που ακούσαμε σήμερα και σας ευχόμαστε καλή δουλειά εντός αυτής της ομάδας, διότι είναι πολύ σημαντική αυτή η δουλειά εντός των πλησίων του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει κύριε Κοχμήριν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξή μας. Και φτάνουμε στις ε, δραστηριότητες που ακολουθούν όσον αφορά την ισότητα των φίλων στις ε, διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Εν συντομία, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για το θέμα. ποια είναι η κατάσταση για την δική μας Επιτροπή αλλά και τις Επιτροπές γενικότερα. Εδώ και μερικές εβδομάδες διεξήχθη μια ακρόαση που ήταν ενδιαφέρουσα και σε αυτή την ακρόαση συζητήσαμε το θέμα των γυναικών και την ένταξή τους στη ζωή και η κυρία Κράτσα μας έστειλε μια έκθεση. Συζητήσαμε επίσης τις γυναίκες επιχειρηματίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης ενδιαφέρον ήταν να δούμε και ποιο είναι το πρόγραμμα της Επιτροπής μας για τον επόμενο χρόνο, η θέση των γυναικών στην πολιτική. Θα είναι έκθεση πρωτοβουλίας που θα έχει συνταχθεί. Μετά θα εξετάσουμε το θέμα των εξωτερικών σχέσεων, τι γίνεται με τις γυναίκες στις περιπτώσεις συγκρούσεων και ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών στις διάφορες ειρηνευτικές ε, διαδικασίες, την εδραίωση της ειρήνης και τον εκδημοκρατισμό. Είναι επίσης σημαντικό να συναντόμαστε με τους βουλευτές που είναι υπεύθυνοι για το θέμα του mainstreaming στις διάφορες επιτροπές δηλαδή της διάστασης των σώτερων στο και θεωρήσαμε ότι ίσως θα πρέπει να ετοιμάσουμε έναν κάποιο κατάλογο με διάφορα θέματα, ένα checklist όπως το αποκαλούμε που θα επιτρέπει την απαρίθμηση διαφόρων πτυχών της ισότητας των φύλων στις διάφορες επιτροπές. Αυτή είναι η πρότασή μας, να καταρτιστεί ένας τέτοιος κατάλογος, checklist, να συμπεριλάβουμε τις διάφορες απόψεις, ούτω ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και το ρετηματολόγιο. Θα είναι ένα εργαλείο που θα είναι χρήσιμο και για την Επιτροπή μας, αλλά και για τις άλλες. οι επιτροπές από τις 21 Σεπτεμβρίου και πέρα υιοθέτησα μια νέα στρατηγική όσον αφορά την ισότητα των φύλων, ε, μια προσέγγιση που θα κρατήσει μέχρι το 2015. Είναι μια στρατηγική που θα συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασιών και θα προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα, ούτως ώστε να υπογραμμίζεται η πτυχή της ισότητας σε όλα τα πολιτικά επίπεδα. Θα ήθελα επίσης εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την ισότητα των φίλων στις διάφορες επιτροπές να λάβουν υπόψη αυτό το κατάλογο, αυτή τη λίστα και να θέτουν ερωτήσεις στους διάφορους επιτρόπους, στους διάφορους πολιτικούς τομείς και να ρωτούν τι έχουν προβλέψει στα προγράμματα εργασιών τους όσον αφορά το θέμα αυτό, ισότητα των φίλων. Είμαστε επίσης υπεύθυνοι για έκθεση πρωτοβουλίας όσον αφορά την διάσταση ισότητας των φύλων στις διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου, το Gender Mainstreaming. Είναι μια έκθεση που θα πρέπει να συντάσσεται κάθε δύο χρόνια και είναι η σειρά μας για το 2011. Θα είναι μια νέα έκθεση πρωτοβουλίας όσον αφορά το θέμα της διάστασης της ισότητας των φύλων, το Gender Mainstreaming. Είναι καλό λοιπόν που θα πρέπει να συντάξουμε αυτή την έκθεση. Είναι σημαντικότατο να επεξεργαστούμε το θέμα και είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο, ερωτηματολόγια τα οποία να μπορούν να συμβουλεύονται διάφοροι υπεύθυνοι για την ισότητα των φίλων στις διάφορες επιτροπές. Θα συμπεριλάβουμε όλα τα σχετικά στοιχεία στην έκθεση πρωτοβουλίας μας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα ερωτηματολόγια αυτά δεν έχουν στο στόχο την υπερφόρτωση του προγράμματος εργασιών των υπευθύνων για το mainstreaming, αντιθέτως θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Θέλουμε να μπορέσουν να κινηθούν βάσει ερωτήσεων που έχουν τεθεί. Η Επιτροπή Ισότητας θα επηρεάσει λοιπόν τις διάφορες επιτροπές και τις εργασίες τους και αυτό από την οπτική γωνία της ισότητας όσον αφορά τα διάφορα πολιτικά ζητήματα. Ξεκινά λοιπόν η συζήτηση. Έχετε εδώ τις ερωτήσεις. Είναι στην ημερήσια διάταξη, τη σημερινή. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας όσον αφορά τον κατάλογο, το checklist και όσον αφορά και το έντυπο. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε επίσης να ακούσουμε και διάφορες προτάσεις γραπτός μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε τον καλύτερο δυνατό κατάλογο με διάφορα σημεία, τον checklist. Και θα μας βοηθήσει στις εργασίες μας κάτι τέτοιο. Δίνω το λόγο στην κυρία Λίχτεμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα την ευκαιρία δυστυχώ να κοιτάξω αυτό το έγγραφο προσεκτικά. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό που έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και γραπτά τις προτάσεις μου. Θέλω να σταθώ σε ένα σημείο μονάχα για το ερωτηματολόγιο. Βλέπω ότι ακριβώς στον τομέα που υπάρχει μεγάλη ε, πρόοδος, ή για θέματα όπου έχουν να κάνουμε τεχνικά θέματα. Βλέπουμε, βλέπουμε πολλές φορές σε τεχνικά θέματα και σε θέματα που προχωρούν ραγδαίως, όπως έλεγα προηγουμένως, στις επιτροπές, στα ακροάσεις να προσκαλούνται σχεδόν αποκλειστικά άνδρες εμπειρογνώμονες. Μπορεί να υπάρχει βέβαια μια κατάσταση, να υπάρχουν καταστάσεις όπου είναι λίγοι οι διεθνείς εμπειρογνώμονες, αλλά όποιος ψάχνει βρίσκει και όλας. Πιστεύω λοιπόν ότι για πάρα πολλά θέματα βλέπουμε μόνο άντρες να έρχονται να μας εξηγήσουν πώς λειτουργεί ο κόσμος και νομίζω ότι και οι γυναίκες γνωρίζουν τα πράγματα αυτά εξίσου καλά. Θα ήταν λοιπόν σημαντικό να δούμε και στο τυπικό αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της πρόσκλησης εμπειρογνώμων να υπάρχει κάποια ισότητα. Να έχουμε λοιπόν μια κάποιος πιο συνδυτή αντιμετώπιση. Να βλέπουμε λοιπόν όταν έχουμε ένα πάνελ από εμπειρογνώμονες να εξασφαλίσετε στο δυνατό βαθμό η ισότητα των φύλων. Γιατί για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Er Σα ευχαριστώ Λίκη πρόεδρο. Ναι, ναι, πράγματι έχει τη Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όπως είπατε κυρία Λίχτενμπεργκερ. Και νομίζω ότι υπάρχει και μία ερώτηση μέσα στο ερωτηματολόγιο. Νομίζω και στο checklist το οποίο είχαμε διατυπώσει είχαμε ζητήσει ακριβώς σε συνεδριάσεις ομάδων εργασίας, σε, σε ακροάσεις εμπειρογνωμόνων, σε ταξίδια αντιπροσωπιών, πάντα να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και η γυναικεία παρουσία. Όπως είπατε πάρα πολλές φορές έχουμε πάνελ που είναι σχεδόν απόλυτα αρσενικά. Και αυτό πολλές φορές συνδέεται με την οικονομική ευρωστία, με την πολιτική εξουσία, με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό που αναφέρατε αυτό το θέμα και θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια πιο έντονη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να υπάρχει και στον τομέα των εμπειρογνωμόνων μια ισότης ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Λίχτεν Μπέργκερ. Κυρία Τόμ. Φωνώ απόλυτα μαζί σας το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τι επιτροπέ αλλά και στα πολιτικά μας κόμματα. Οργανώνουμε ακροάσεις μόνο με ε, άντρες ομιλητές. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να τα δούμε πολλά θέματα ε, από τη σκοπιά της ισότητας των δύο φύλων και μπορούμε να εισάγουμε το θέμα της ισότητας των δύο φύλων σε πολλούς άλλους τομείς που δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα ας πούμε, ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική ε, δημιουργίας θέσης απασχόλησης για να ε, διορθώσουμε την αγορά εργασίας που καταδυναστεύεται, αν θέλετε, από τους άνδρες. Σε όλα τα θέματα με τα οποία ασχολούμεθα θα πρέπει να έχουμε κατά νου την διάσταση της ισότητας των δύο φύλων. Μέχρι τώρα δεν γινόταν κάτι τέτοιο. Το προσπαθούμε να το μάθουμε ε, και είναι δύσκολο. Είναι μια μεγάλη διαδικασία και απαιτεί πολλή δουλειά στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σε άλλες και σε άλλες πολλές επιτροπές όπου θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό το θέμα, αυτή η διάσταση της ισότητας των δύο φίλων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόμψον. Κοιτάξτε, πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να βελτιώνουμε την, τα θέματα ισότητας. Ακούγοντάς σας, σκέφτομαι ότι στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, οργανώθηκε μια συνάντηση πρωθυπουργών, σημαντική συνάντηση, και όταν ο Πρωθυπουργό μας πήρε το πρόγραμμα, είδε ότι σαν εμπειρογνώμονες είχαν προσπιθεί μόνο άντρες και πραγματικά πήρε μια ριζοσπαστική απόφαση θεώρησε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν σωστό, εξού και μποϊκόταρε τη συνάντηση. Δεν πήγε είναι λίγο υπερβολική σαν αντίδραση θα έλεγα, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιοι που, το, ε, που ασχολούνται αν θέλετε, που τους ενδιαφέρει το θέμα αυτό της ισότητας. Και νομίζω ότι και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας, γιατί ήρθατε εδώ να συζητήσουμε. Θα ξαναβρεθούμε βέβαια σαν υπεύθυνε για το gender mainstreaming και περιμένω την, τις απόψεις σας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Τώρα, στις 4.30 θα αρχίζει ε, η συνεδρία της Επιτροπής. 4.30.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 Eh, Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να χαιρετήσω καταρχάς ε, τους βουλευτές, ε, την φιλοξενούμενή μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σε αυτή την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την ε, Επιτροπή Ισότητας. εδώ και 10 χρόνια καταλήξαμε στην 1325, στο ψήφισμα 13.125 που αφορά την αντιμετώπιση των γυναικών σε περιόδους κρίσεων, σε περιόδους πολέμων και ε, ασχοληθήκαμε με τις εμπειρίες των γυναικών, με την ε, συνεισφορά των γυναικών στην ε, επίλυση, στις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων και την ειρηνευτική διαδικασία εν γέννη. Θελήσαμε να συνεδριάσουμε από κοινού με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ε, θέλουμε όλοι να συνεργαστούμε μέσα στα πλαίσια του ψηφίσματος 1325. Πρόκειται για μια κοινή συνεδρίαση όπως σας είπα, επομένως έχουμε δύο προέδρους. Θα συμπροεδρεύσουμε σήμερα το απόγευμα. Θα δώσω το λόγο την κυρία Χαουταλά, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η κυρία Χάουταλα. Έχουμε συζητήσει, συζητήσαμε μακρόν στην Επιτροπή ε, τα προβλήματα που απασχολούν το Μεξικό. Γι' αυτό δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω εν γέρος. Καθυστέρησα λίγο ε, για λόγους που δεν μπορούσα να ελέγξω. Λοιπόν, ε, κάτω από διάφορες συνθήκες κατα καταφέραμε να κάνουμε να λειτουργήσει το ψήφισμα τα τελευταία 10 χρόνια, το 1325. Στην Φιλανδία συνεργάστηκα πάρα πολύ στενά με την κυρία Elizabeth Ρέινε, η οποία ε, συνεργάζεται και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Και και με την κυρία Helen Charlie Johnson, την πρόεδρο της Λιβερίας ο ΙΕ αντιμετωπίζει πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα που αφορούν τον ρόλο των γυναικών σε περιπτώσεις συγκρούσεων, διότι οι γυναίκες είναι θύματα μεν αυτών των συγκρούσεων, όμως μπορούν ταυτόχρονα να επηρεάσουν τις εξελίξεις και να συνεισφέρουν στην επίλυση των προβλημάτων ή τουλάχιστον μπορούν να συνεισφέρουν στην σταθεροποίηση της κατάστασης. Μετά την μελέτη ε, που έχουν γίνει, μετά ε, την μελέτη των ε, εξελίξεων, βλέπουμε ποια είναι η γενικότερη και, μπορούμε να δούμε ποιες, ποιες είναι και οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και ε, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και εμείς και τα όσα έχουν αποφασιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, θα πρέπει δηλαδή ούτως ή άλλως τα αποτελέσματα του 1325 να ενσωματωθούν στην νομοθεσία μας. Λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματα στο οποίο έχουμε καταλήξει. Ότι καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει ένας κωδικός ε, αντιμετώπισης συμπεριφοράς, θα πρέπει να δοθούν κάποια κονδύλια για τα θέματα ισότητας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει ε, τη συνεργασία της με τους τοπικούς οργανισμούς, με τοπικούς φορείς, ε, με, τη, με τους υπεύθυνους για την απόκτηση προσόντων, κυρίως, κυρίως επαγγελματικών προσόντων από των γυναικών. Η κατευθυντήρια γραμμή, αν θέλετε, στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια συνεκτική αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του ψηφίσματος ε, του ΟΗΕ για το 1325 ε, και του ψηφίσματος που αφορά την σταθερότητα και την ειρήνη. Το 2008 το Δεκέμβριο υιοθετήθηκαν, το τελευταίο αυτό κείμενο για να, και ρυθμίζει μάλλον τις ενέργειες και τις δράσεις των διαφόρων επιμέρους φορέων που δρούν σε τοπικό επίπεδο, π.χ. στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η... Αποφασίσαμε να δημιουργήσουν, αποφάσισε ο ΙΕ να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο οργανισμό που αφορά, με συγκεκριμένη υπηρεσία που αφορά τις γυναίκες ιστορικής σημασίας και ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό οι γυναίκες θα ταχθούν καλύτερα στις δραστηριότητες και στην δομή του ΟΗΕ. Είδαμε ότι η κυρία Μπασελέ, η κυρία Μισελ Μπασελέ, η πρώην πρόεδρος της Χιλής, διορίστηκε ε, σαν εκτελεστική διευθύντρια κάτω ακριβώς από τον Γενικό Γραμματεία του ΟΗΕ και θα αναλάβει δράση από το 2011 για τον ΟΗΕ των γυναικών. Στο Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου του 2009 υιοθετήθηκε ε, ένα ψήφισμα για την, που αφορούσε την ε, σεξουαλική βία. Είδαμε ότι δημιουργήθηκε και διορίστηκε ένας ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που αφορά την ε, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, που θα ασχολείται με τα θέματα σεξουαλικής ε, ε, κακοποίησης των παιδιών. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Το Φεβρουάριο του 2010 τη θέση αυτή ανέλαβε η πρώην Επίτροπος η κυρία Βάλστρομα και γνωρίζοντας την κυρία Βάλστρομα και το πόσο δυνατή είναι πιστεύω ότι θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες Τη θέση αυτής. Ε, ή είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται ε, να κλείσει τα μάτια και στα θέματα ε, της βίας κατά των γυναικών που είναι θέμα το σχετικό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασχοληθεί ακόμα περισσότερα ε, με τα θέματα ισότητας των δύο φύλων και σε όλες τις εξωτερικές δράσεις μας. Είδαμε ότι το 35% των, ε, της αναπτυξιακής βοήθειας της Κομισιόν ε, δαπανάται σε σχέδια τα οποία έχουν μια σημαντική πτυχή ισότητας των δύο φύλων Ήδη υπάρχει μια πρόεδρος, πρόοδος σημαντική. Ο κύριος Άτι ε, ο πρώην πρόεδρος της ε, Φιλανδίας, ε, όταν δραστηριοποιείται για τα θέματα διαμεσολάβησης για την ειρήνη όταν ήταν διαμεσολαβητής και πήγαινε σε μια συνάντηση πάντα ρωτούσε που είναι οι γυναίκες ε, όταν συναντούσε μονάχα άντρες. Λοιπόν, ούτως ή άλλως έχουν γίνει διάφορες δηλώσεις, ε, διάφορα ψηφίσματα έχουν υιοθετηθεί ε, με βάση το ψήφισμα του 1325. Το Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει διάφορα κείμενα σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων. Υπάρχει μια συνεκτική κοινοτική αντιμετώπιση για το ψήφισμα 1425 και 8120. Επίσης ε, υπάρχει η χάρτα για τα δικαιώματα των γυναικών, τα οποία επέβαλε η κυρία Ρέντινγκ. Και ε, θα ήθελα να δώσω την, ε, τον λόγο στην ομιλήτριά μας, την κυρία Γκία, για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που ανέθεσε αυτή τη σημαντικότητα τη μελέτη. Στόχος της μελέτης ήταν να έχουμε μία βάση των πάντων με γενική έποψη όσον αφορά το 1325, τον 1820 και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο το φάσμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά και τις γυναίκες στις ένοπλες σειράξεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ εκείνους που με βοήθησαν στην διεξαγωγή της μελέτης, προσωπικό της ΆΙΖΑΣ Ευρώπη, τον Φρανσίσκο Πενάλβα και τον Σεμβάστιαν Μπλόκιν και, Κύριε Κράτσα, επίση που βοήθησε στο πρώτο τμήμα. Έρχεται να αντιγραφώ, δεν θα διατρέξω τις 180 σελίδες. Οι μισές είναι παράρτημα, αλλά θα αναφερθώ στα βασικά σημεία, τα βασικά πορίσματα και πιο σημαντικά τις διάφορες συστάσεις σχετικά με την πορεία, τη μελλοντική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πώς μπορεί να βοηθήσει το Κοινοβούλιο. θέλω να πω ότι η έρευνα έγινε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο του 2010, άρα υπάρχει ένα εξάμεινο κενό Εν τω μεταξύ ίσως να υπήρξαν εξελίξεις, ίσως και όχι. Αυτή η μελέτη θα δημοσιευθεί το Νοέμβριο. Υπάρχουν και άλλοι υπέροχοι εδώ, οι δήμονες που μπορούν να σχολιάσουν, αφού θα αναφερθώ εγώ στην έκθεση. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορη. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερες ερωτήσεις για να απαντήσω, γιατί το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε όλοι στο σπίτι σας εξάλλου. Αναφερόμενοι λοιπόν σε αυτά που είπε η Χάιντι, να δούμε αν λειτουργεί έξοχα. Λοιπόν, Κάτι λείπει. While I talk, if you can just give me minutes. Άμα επιτρέψετε ένα πεντάλεπτο, διότι εδώ είναι λάθος η παρουσίαση στον υπολογιστή διαφάνειας. Μισό λεπτό. Φόρτωσα τη λάθο παρουσίαση γιατί την είχα την άλλη σε διαφορετικό υπολογιστή. Λοιπόν, θα αναφερθώ στους βασικές προδιαγραφές. Θέλαμε να δούμε τα επιτέγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που ήθελε το Κοινοβούλιο να κάνουμε είναι αυτό να το πλαισιώσουμε. Σχετικά με αυτά που έκανε και ο ίδιος η ΕΤ τελευταία δέκα χρόνια, διότι Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι μέλη του ΟΗΕ και οι 1325 και οι 1820 και διάφορες σχετικές, ε, τα σχετικά ψηφίσματα αφορούν το πώς μπορούμε να προωθήσουμε προσπάθειες κατά της βίας εναντίον των γυναικών σε συγκρούσεις. Και έγινε μια μελέτη το 2009 για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που εμπερίχει περισσότερες πτυχέ σχετικά με το gender mainstreaming στο Κοινοβούλιο και στις εξωτερικέ σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ωραία, εκτόξευση. Ζητώ συγγνώμη. Α, αυτό ήθελα, ωραία. Λοιπόν, αυτά που είπε η Χάιντι συνεχίζουμε εδώ και υπάρχει μια καλή συνέχεια πηγαίνοντα από τον ΟΗΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ότι ξέρουμε η Μάργκο Βάλστρομ είναι η ειδική εκπρόσωπο, αντιπρόσωπο, ήταν τα δυναμική το τελευταίο εξάμεινο. Έχω αυτή την παράθεση γιατί έτσι αισθάνομαι εγώ σχετικά με τα, εκεί, τα σημεία που ιστορούμε. Έγινε μια, έκανα μια ε, συνειδητή προσπάθεια να σταματήσω να επαναλαμβάνω. Είναι τόσο περίπλοκο, τόσο δύσκολο. Εάν μπορούμε να απαγορεύσουμε τι βόμβε διασπορά, γιατί δεν μπορούμε να, μπορούμε να απαγορεύσουμε και την σεξουαλική βία στι συγκρούσει, στι σειράξει. Θα ήθελα εδώ να σας δείξω αυτό που βλέπετε σε σελίδα 5 της ε, μελέτης. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες ως αριθμούς, τις γυναίκες ως θύματα, αλλά τις γυναίκες ως δημοσιολαβήτριες, σαν φορείς αλλαγής και στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ενώσεως εδώ μπροστά σας βλέπετε τρεις πτυχές. Έχουμε τη διπλωματική δράση, όπου έχουμε την ύπατη εκπρόσωπο, έχουμε μια γυναίκα εκεί, επιτέλους, ε, τη Ρώσαλιν Μάζνομ για το Σουδάν. Έχουμε πολυμερείς ε, διμερέη προγραμματισμό, διαχείριση του, των κρίσεων και στο πλαίσιο που έχουμε μετά την Λισαβόνα δημιουργείται η, Ευρωπαϊκή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ποιος εργάζεται πού. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που σε αυτό το τομέα των εξωτερικών σχέσεων έχει βελτιωθεί η θέση του, ε, είναι συμβουλευτική εξουσία που έχει το Κοινοβούλιο και βέβαια υπάρχει και η εξουσία που έχει το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον προπολογισμό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να μιλήσουμε λοιπόν και τη διμερή δουλειά που κάνουν τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παίρνει και δύναμη και από τη δουλειά που γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών και από τη προσπάθεια. Πάμε τώρα στι προδιαγραφέ. Λοιπόν, τι αναλύσαμε. Τη γενική προσέγγιση που αναφέρθηκε και την τριπλή προσέγγιση που εφαρμόστηκε επί Γαλλικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως που εξέτασε την πολιτικό διάλογο, διάλογο πολιτικής, την ε, προσέγγιση όσον αφορά τη συμπερίληψη της διάστασης των φύλων ε, στις διάφορες πολιτικές και υποστήριξη διαφόρων στατηγικών δράσεων και έχουμε τις δύο δράσεις η IDHR και IFS και όσον αφορά τις έναπλες σειράξεις πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ασχοληθούμε να εφαρμόσουμε ε, τα ψηφίσματα και μετά έχουμε και τι κατευθύνσει γραμμέ Ευρωπαϊκή Ενώσεω στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Επί υπάρχουν επιρέστατα παρατήματα όπου το προσωπικό που συνεργάστηκε μαζί μου ε, έκανε σύγκριση, κάναμε σύγκριση όλων των εγγράφων, οπότε είναι η πρώτη βάση δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει, δεν θα τα αναφέρω όλα, βλέπετε μια συγκριτική εικόνα ε, τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτά που έκανε ε, το ΙΕ 1325. Λοιπόν, μεθοδολογία, εξετάσαμε την τεκμηρίωση, δεν υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα, αυτό ήταν και ο λόγος ύπαρξης μελέτης. Κάναμε συνεντεύξεις με τους βασικούς παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τέσσερα χρόνια εργάστηκα στις Βρυξέλλες και ξέρω τους πιο σημαντικούς ανθρώπους εδώ. εμπειρία από αποστολές, πήγα στις διάφορες αποστολές. Ε, είναι μιλάμε ο ένας με τον άλλον όσον αφορά την κοινότητα για την ισότητα των φύλων, οπότε έχουμε πάρα πολύ καλέ πληροφορίε. και κάναμε ποιοτική και ποσοτική στατιστική ανάλυση. Εξετάσαμε όλες τις κοινέ δράσει των αποστολών τη ΚΕΠΑ. Ε, ήταν σαν να εξετάσαμε τι γίνεται ελληνευτικέ επιχειρήσεις και θέλαμε να δούμε τι συμπεριλαμβάνει πώ αναφέρονται τα ανθρώπινα, πώ συζητιώ τα ανθρώπινα δικαιώματα στι 1325 και με ποιο τρόπο αναλύσαμε το προσωπικό που εργάζεται για την εφαρμογή την 1325 και κάναμε ανάλυση των κονδυλίων και των οικονομικών μέσων που διατίθενται για την επιτύχηση του σκοπού. Λοιπόν, το βασικό θέμα, η βασική διαφορά, τα κενά που διαπιστώσαμε, ποια ήταν. Βασική διαφορά αναφέρεται πολύ σωστά στο παράτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών τη Ευρωπαϊκή Ενώση για τη βία κατά των γυναικών. Και αυτό τονίζουμε εδώ. Η πολιτική σταθή και ένοπλε συγκρούσει ξέρουμε ότι δημιουργούν ανισορροπίε. Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στους αφατήτες της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Διαδίδονται πάρα πολύ ε, τα όπλα και αυτό οδηγεί σε βία και παρά αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνδέει τους διάφορους τομείς τη στρατηγικής μέχρι τώρα. Είχαμε ε, την την ανάπτυξη στρατηγική δεν συνδέσει και το θέμα τη ότητας των φίλων και τη γη κατά των γυναικών μάλλον με τα όπλα. Και τι γίνεται και κυρίως και τι, ποιες είναι οι συνέπειε και τη ε, βία ε, στο σπίτι. Οι εξελίξει στον ΟΗΕ, για εσά που δεν γνωρίζετε το τομέα, τα τελευταία χρόνια, δέκα χρόνια πέρασαν, είναι γελίο που χρειάστηκε τόσο χρόνο για να εφαρμόσουμε πραγματικέ δράσεις. Έχουμε δείκτες του ΟΗΕ, θα αναφερθούμε σε αυτό αργότερα. Υπάρχει σχέδιο δράση του ΟΗΕ για όλο τον ΙΕ παρά τον 1325 που προωθεί και ενθαρρύνει τη δημιουργία εθνικών σχεδίων δράσης για το 1325 δεν υπήρχαν κάποια πλαίσια και κατευθύνες γραμμές και δεν υπάρχει σαφής προσανατολισμός. Πρόσφατα έχουμε σχέδια δράση. Ο διορισμός βεβαίως της κυρίας Βάλστρομ βοήθησε Ντάγκ μπορεί το παρακαλώ λίγο. Η Μάργκο Βάστρομ ε, έκανε μια πολύ έγκαιρη μελέτη, σημαντική έκανε ανάλυση των πρακτικών που ακολουθούνται όσον αφορά την ε, πρόθεση της ειρήνης και διατήρηση της ειρήνης και είναι πολύ καλό οδηγό που μπορούσε να χρησιμοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ε, δράσεις της. Κοιτάμε ε, όλες τις πτυχές τις εμπεριλαμβάνουμε και δίνουμε πληροφορίες που είναι χρήσιμες για, τους, για όλους που πρέπει να εφαρμόσουν επιτόπου τις δράσεις. Αυτό το κενό είχαμε πριν. Να βοηθήσουμε εκείνους που επιτόπου να εφαρμόσουν τις δράσεις. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, πρέπει να το εξετάσουν όλοι. Βεβαίως, πρόθεση εθνικών σχεδίων δράσης. Είχαμε αρκετά το τελευταίο χρόνο. Πάρα πολύ σημαντικό και σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ να συνεργάζονται Έχουμε την συνεργασία για την ισότητα των φύλων και ανάπτυξη που κράτησε μερικά χρόνια και έχουμε μια αναθεώρηση του 2010 που δεν ήταν έτοιμη εγκαίρω για τη δική μα μελέτη. Κάτι άλλο πρέπει να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να αντλήσει κάποια μαθήματα. Λοιπόν, ε, έχουμε νομικά δεσμευτικέ στοιχείε. οι γυναίκε έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε διάφορου τομεί, Η βία κατά των γυναικών τώρα γίνονται πολλές προσπάθειες στον τομέα και τώρα αναφέρουμε στο καθετικό της Ρώμης ότι είναι παραδίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά από 10 χρόνια και ακόμα έχουμε περισσότερες αποτυχίες από ό,τι επιτυχίες. <coughs> Λοιπόν, αυτό που είδαμε δεν είναι μόνο στη μελέτη, αλλά το επαναλαμβάνει η μελέτη, αυτό που λένε όλοι επαναλαμβάνει η μελέτη. Πέραν από τους θεσμούς, οι μη κυβερνικέ οργανώσει και τα δίκτυα των γυναικών είναι η βασική φορεί των αλλαγών. Και όπω είπε η Χάιντι, θα πρέπει να εξακολουθούμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση, όχι μόνο να ενθαρρύνουμε και να λέμε ότι θα υπάρξει διάλογο, αλλά πρέπει να δούμε και ποιε είναι οι επίσημε δομέ που υπάρχουν στι χώρε μα. Η αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο εκεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το σχηροποιήσει αυτό μέσω τη υποστήριξη με χρήματα. Και εδώ το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το πλαίσιο πολιτική που ακολουθεί που είναι ad hoc προσεγγίσεις, όπως είναι οι περισσότερες προσπάσεις... στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσης, να υποστηρίξει και να εφαρμόσει το 1325 και τις, α, ε, τα άλλα ψηφίσματα. Βασικά και ένα έλλειψη ηγεσίας της Ευρωπαϊκής θα αναφερθώ σε αυτό σε λίγο, έλλειψη σημαντικής εφαρμογής, έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών. Και τώρα βλέπετε εδώ, και επαναλαμβάνω αυτό, τα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά καλά, κυρίως ε, ένα από τα πράγματα που μας ζητήθηκε να αναλύσουμε εξέταζε την εφαρμογή τη 1325 και τη 1820 στις αποστολές της ΚΕΠΑ και είναι ένα πάρα πολύ καλό έγγραφο για κατεύθυνση. Δεν το εφαρμόζουν όμως. Γιατί? Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο άτομο για την εφαρμογή αυτών. Και αυτό είναι απλούστατο. Τόσο απλό είναι. Και το ίδιο ισχύει και τα περισσότερα άλλα έγγραφα. Παρόλο που υπάρχουν κάπω περισσότερε Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη, υπάρχουν πολύ περισσότερο για την κοινωνική απασχόληση, αλλά θα πρέπει το την, τα εσωτερικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ενώσης να συνδέσουμε τα εξωτερικά. Πρέπει να υπάρξει μια τέτοια γεφύρωση λοιπόν. Λοιπόν, εσωτερικά έγγραφα είναι ο δικός χάρτης για την ισότητα που πρέπει και να θεωρηθεί φέτος νομίζω. Η εντολή για την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρόγραμμα Δάφνη που ήταν επιτυχέστατο. Να μην ξεχνάτε ότι και αυτό εξετάζει το θέμα της βίας κατά των γυναικών στις συγκρούσεις, στις ένοπλες και πάντα και στην, ε, στο εμπόριο γυναικών και στο εμπόριο γυναικών υπάρχει και σχετισμός με τα όπλα. Υπάρχουν πολλά πορίσματα. Ποια είναι τα όρια της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει. Θα αναφερθώ στο θέμα αυτό. Βρήκαμε ότι υπάρχει φραδίτη στην ε, αντιμετώπιση, υπάρχει έλλειψη ταχείας προειδοποίησης. Το θέμα των εντολών για τις αποστολές που δεν έχουν συγκεκριμένες κατευθυντικές γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη 1325. Δεν υπάρχουν κίνητα για να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου. ανθρώπινα δικαιώματα υποτίθεται ότι έχουν ήδη ενσωματωθεί. Και φυσικά το θέμα είναι ποιο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή τη διάσταση του φύλου. Ο καθένα νομίζει ότι είναι κάποιο άλλο. Υπάρχει μία γυναίκα για δείγμα πάντα που υποτίθεται ότι αυτή είναι η αρμόδια σε αυτόν τον τομέα. Η εφαρμογή λοιπόν όλα αυτά είναι ακόμα ad hoc μέσα στα πλαίσια του πλαισίου EAS. Η μονάδα της ειδικής ε, ε, αντιπροσώπου τώρα έχει ενσωματωθεί στο EAS. Δεν έχει πια ε, μια σαφή θέση και χρειάζεται να υπάρξει πίεση για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα ισχυρό τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα λοιπόν είναι ποιο είναι αρμόδιο. Σε πολλέ περιπτώσει δεν υπάρχει η κατάλληλη λοιπόν αρχιτεκτονική και δεν έχουμε και του απαραίτητου πόρου. Οικονομικού είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για την εφαρμογή του 1325 του ψηφίσματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά <clears throat> αυτό είναι πάρεργο για αυτούς. Είναι ένα τμήμα της συνολικής τους δραστηριότητας, αλλά είναι ίσως το 10% της δραστηριότητάς Πρέπει να υπάρξει κατάλληλη εστίαση και κατάλληλη προσπάθεια στον τομέα αυτό. Η κυρία Άστον αυτή τη στιγμή κυρίως ενδιαφέρεται να προωθήσει το λεγόμενο gender mainstream, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Δεν λέω ότι αυτό είναι απρόσημα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ενσωματώσει κανείς αυτή τη διάσταση αν δεν υπάρχει η κατάλληλη αρχιτεκτονική και δεν υπάρχουν σημεία αναφοράς. Ίσως ο ΙΕ <clears throat> μπορεί να δράσει μέσω της οργάνωσης αυτής για, τον, για τις γυναίκες στον ΟΗΕ, αλλά είναι πρόωρο να κάνει κανείς μια τέτοια πολιτική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, αν δεν έχει ήδη την κατάλληλη αρχιτεκτονική. Και φυσικά υπάρχουν και τα θέματα βελτίστων πρακτικών που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτό το οποίο θα σας πω όμως είναι ότι υπήρξαν και μερικά θετικά στοιχεία, ιδίως τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουμε τους εμπειρογνώμονες που είναι πολλές φορές νεαρές κοπέλες στα κράτη-μέλη. Τώρα έχουμε προχωρήσει αυτή την αρχική αντιμετώπιση σε μια πρόσφατη συνεδρίαση σε ψηλό επίπεδο, σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν επιτευχθεί λοιπόν πολλά τα τελευταία πέντε χρόνια. Πολύ καλές πρωτοβουλίες, αλλά είναι άτυπες, είναι ανεπίσημες. Η ομάδα κρούσης λοιπόν, που είναι από τα ίδια μέλη που βρίσκονται στα κράτη-μέλη, κάνουν <clears throat> καλά πράγματα, αλλά υπάρχει και πρόβλημα με, το, με τις προσωπικότητες των ατόμων αυτών. Υπάρχουν επίσης τα άτομα τα οποία είναι οι αιστείες των δραστηριοτήτων για, τα, για το φύλλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάπου μια καμιά τρακοσαριά άτομα εργάζονται για τα θέματα αυτά. Αλλά πολύ λίγοι από αυτούς έχουν πλήρη απασχόληση. Ίσως είναι καμιά δεκαριά το πολύ οι άνθρωποι που δουλεύουν σε πλήρη βάση. Υπάρχει ένα δίκτυο εστιακών σημείων, το AIDCO το οποίο είναι πολύ καλό για να αποσπά πληροφορίες και έχουν μια πολύ καλή εσωτερική δομή. Και έχει φύγει αυτός ο οποίος δούλευε το εσωτερικό τους διαδίκτυο, το ίντρανέτ Αυτό σημαίνει λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν πολύ καλά σε ανεπίσημο επίπεδο, αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο γιατί δεν υπάρχει μια πιο επισημοποιημένη δομή. Κοινέ δράσει. Υπάρχουν τώρα περισσότεροι εμπειρογνώμες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχει περισσότερη ε, ανταλλαγή καλών αλλά και κακών πρακτικών. Πέρσι έγιναν κάποιες ε, ε, συναντήσεις με συμβούλους για θέματα φύλου και υπάρχει και ένας ε, τέτοιος εμπειρογνώμος σε κάθε αποστολή εκτός από τη Γουινέα Μπισάου. Και γίνονται προσπάθειες επίσης για καλύτερη εκπαίδευση, ιδίω στις αποστολές της ΚΕΠΑ κτλ. Αλλά δεν έχουμε ακόμα τυποποίηση και εναρμόνιση. Γιατί όλα αυτά τα θέματα αποφασίζονται από τα κράτη-μέλη τι ομάδε θα αναπτύξουν, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσει την τυποποίηση και την εναρμόνιση για αυτή την εκπαίδευση. Η Σλοβενική Προεδρία είχε δημιουργήσει και ένα ενεχειρίδιο το οποίο περιλάμβανε όλες αυτές τις πολιτικές και τις είχε συμπηλήσει, αλλά θα πρέπει να τις ξανά εκ νέου συμπηλήσουμε γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έχουμε επιτέλους και κάποιους δείκτες, στους οποίους θα έρθω τώρα, και υπάρχουν και οι ομάδες ε, κρούσης και οι πλατφόρμες των μη κυβερνητικών οργανώσεων που υποστηρίζουν σχέδια δράσης και επίσης όλα αυτά γίνονται στις χώρες όπου υπάρχει βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκλήσεις εδώ εκ νέου επαναλαμβάνουμε. Χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται μια τέτοια στρατηγική για το φύλλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εάν δεν υπάρχει δομή, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε πόρους. Αυτό είναι η λεγόμενη παγίδα του ΚΑΤΣ 22. Πως σε πολλά κρατημέλη δεν υπάρχουν εθνικά σχέδια δράσης γιατί δεν θεωρούν να απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει όμως να έχουμε εναρμονισμένες προσεγγίσεις και θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνοντας ένα γενικό κατευθυντήριο πλαίσιο για εναρμόνιση. Φάνηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φάνηκε και από το ΝΑΤΟ ότι δεν έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει το πλαίσιο αυτό να ενδυναμωθεί. Λοιπόν, ας δούμε τώρα ε, τους μακροπρόθεσμους ε, στόχους και συνδέσμους. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τοπικούς παράγοντες, ε, προφανώς. Απ' την άλλη πλευρά το θέμα είναι ποιος είναι υπόλογος, πώς ελέγχεται το όλο σύστημα. Δεν, δεν μπορείτε να τα δείτε αυτά, γιατί υπάρχει, υπάρχουν όμως το κείμενο. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι υπάρχουν δείκτες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εφαρμόσει μια ολόκληρη διαδικασία. Ε, μην ξεχνάμε ότι το θέμα μας είναι οι, μελέτη, γυναίκες ε, και η μελέτη των γυναικών στα θέματα ενόπλων συγκρούσεων. Λοιπόν, στους δείκτες εδώ έχουμε αριθμητικούς δείκτες, ε, τα ποσοστά γυναικών ε, που έχουν ειδικέ γνώσεις, ε, συνεργασία σε προγράμματα εκπαιδευτικά, αναλογίες και ποσοστά ανδρών και γυναικών, πρόσφυγες, μετανάστες κτλ. Αυτοί είναι προτινόμενοι δείκτες ε, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας που ασχολήθηκε λίγο με τα θέματα των γυναικών και ένοπλων ε, σειράξεων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούμε λίγο δύο παράλληλες ε, πορείες γιατί δεν έχουμε δείκτες ε, που να αφορούν ε, αποκλειστικά και μόνο τις γυναίκες σε, ένοπλες, σε περιόδους ένοπλων σειράξεων, εκτός από τους δείκτες που ισχύουν στις χώρες που εφαρμόζουν το 1325. Θέλετε να ολοκληρώσω, ε? Ωραία. Τρεις διαφάνειες έχω ακόμα. Ένα τελευταίο σχόλιο. Όλα όλοι, όλα, τα, όλα τα κονδύλια και όλα, όλοι οι πόροι έχουν αναφορές στα θέματα του, της ισότητας των δύο φύλων του 13-25, όχι όμως σαφ, σαφώς, δεν εμφανίζονται σαφώς. Και η ομάδα υψηλού επίπεδου θεωρεί ότι μπορεί να υποστηρίξει την εργασία της άτυπης ομάδας κρούσης για τις κατευθυντές γραμμές. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι απόλυτα ανοιχτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω και το Κοινοβούλιο μπορεί να γίνει πολιτικός καταλήτης για την πρόοδο των θεμάτων. Αρχίσουμε λοιπόν την συζήτηση. Είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε να λάβετε το λόγο και να θέσετε ερωτήματα. Η κυρία Λούνα Τσεκ. Ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές ε, πληροφορίες σχετικά με τα επιτεύγματα και τα κενά που υπάρχουν. Πριν από δύο μήνες ήμουνα σε μια συνάντηση περιφερειακή για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνάντηση των Λόμπι, όπου μέλη της UNIFEM Νέας Υόρκης παρουσίασαν τα προβλήματα. Ήταν παρόμοια εικόνα. Ίσως και χειρότερη από αυτή που παρουσίασατε εσείς υπήρχαν έγγραφα, υπάρχουν σχέδια δράσης, προθυμία, λείπει εφαρμογή και τα χρήματα. Και οι γυναίκες σε υψηλέ θέσεις. Υπάρχει μικρή βελτίωση στη δεκαετία, αλλά δεν αρκεί αυτό. Όπως είπατε, το ίδιο έλλειψη ηγεσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προβλήματα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ταυτίζεται με αυτά που συζητούσαμε κι εμείς. Αυτά που είπαμε στην Κάθριν Άστον. Διότι όπως είπατε είναι πολύ ισχυρή όσον αφορά το mainstreaming. Θέλει το mainstreaming. Αλλά είναι και το θέμα ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα των φύλων. Αν δεν υπάρχει σωστή δομή, πώ θα γίνει το mainstreaming σε αυτό το τομέα. Να ρωτήσω κάτι για το Ulex, γιατί είμαι συγγήτρια του Κοινοβουλίου για το Κωσυφοπαίδιο. Και συναντήθηκα επανειλημμένα. Με τον παλιό στρατηγό του Ulex και το προσωπικό του. πώς κρίνεται τη δουλειά τους για τα θέματα ισότητας των φύλων. Και εντός γιούλεξ και προβολή προς τα έξω. Ευχαριστώ που είπατε ότι τα δίκτυα μη κυβερνητικών οργανώσεων των γυναικών είναι εκείνα που προωθούν το θέμα μας. Χρειαζόμαστε τους φορείς της μη κυβερνητικές οργανώσεων των γυναικών για να ασκήσουν πιέσεις δεν αρκούν μόνο αυτά που κάνουμε εμεί. Σαν μέλο του Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή ΣΕΔ και στην ΑΦΕΤ, πρέπει να κάνουμε δουλειά εμεί. Τα προεδρία τη ΑΦΕΤ ΣΕΔ είναι αποκλειστικά από άντρε αποτελούνται. Και στι αντιπροσωπείε που έχουμε στον κόσμο, μόνο δύο αυτών ηγούνται γυναίκε. Των υπολείπων ηγούνται άντρε. Πρέπει να κάνουμε πολλά για να βελτιώσουμε την ορατότητα των γυναικών σε υψηλό επίπεδο, κυρίω σε διεθνεί υποθέσει. Ήμουν συνεδρίαση στο Εκουαδόρ τη Eurolat και συζήτηση για την άμυνα και την ασφάλεια. Μόνο εγώ και μία άλλη εκπρόσωπο γυναίκα από τι χώρε Λατινική Αμερική μίλησαν. Άρα πρέπει να κάνουμε περισσότερο όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Τζιπ, τον αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμμετέχει στη συζήτηση για τα θέματα της ισότητας. Η κυρία Ντεμπρούν και μετά η κυρία Μπραντνερ, οι επόμενοι θα πάρουν το λόγο. Κυρία Ντεμπρούν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είπε η κυρία Αγγία ότι είχε εξετάσει ορισμένα από τα εσωτερικά προγράμματα, ατενίζον ιδιαίτερα τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Αναρωτιέμαι αν έχετε κοιτάξει το ειδικό πρόγραμμα ειρήνης και συμφιλίωσης του ΟΗΕ για την Ιρλανδία. Αυτό είναι ένα εσωτερικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε, αλλά είχε ακριβώς να αντιμετωπίσει καταστάσεις αντιπαράθεσης και σύγκρουσης και εξόδου από τη σύγκρουση αυτή. Υπήρχαν τρία τέτοια προγράμματα, το PIS 1, PIS 2, PIS 3, δηλαδή ειρήνη 1, 2, 3 και είχαν και κάποια ειδικά προγράμματα για τις γυναίκες. Μπορεί αυτό να μην, σας, να μην το θεωρήσετε ότι είναι διαφορετικό, αλλά για μένα νομίζω ότι μπορεί να έχει θετικά στοιχεία. <clears throat> Εγώ πριν έρθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα, είχα εμπλεκεί, εμπλακεί συγγνώμη, και στις ε, διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην Συμφωνία για την Ειρήνευση στην Βόρεια Ιρλανδία και τον Belfast και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς μια συνεχή παρακολούθηση και να εξασφαλίσει ότι οι γυναίκες συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και να αναγνωρίζει το ρόλο των γυναικών στην οικοδόμηση ειρήνη και τη συμφιλίωση. Γιατί χωρί τι γυναίκε, και αν οι ίδιοι οι διαπραγματεύτε δεν έχουν επίγνωση αυτού του θέματο, απλώ επαναλαμβάνεται και ανανεώνεται η ίδια κατάσταση ε, αντιπαράθεση. Κύριε Μπράντρε τώρα, σας ευχαριστώ Ζιέζη για αυτή την έκθεση είναι παράξενο όταν μιλάει κανείς για τα έγγραφα αυτά του 2008. Φαίνεται να είναι πολύ παλιό αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτή η έκθεση έχει θέτει ένα βασικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ καλό. Θεωρούσατε ότι τώρα ήταν πιο εύκολο να έχει κανείς πρόσβαση στις διάφορες προσωπικότητες και να βλέπει τι γίνεται από ότι στο παρελθόν πριν από δύο-τρία χρόνια. Θυμάμαι ότι είχε συνεργαστεί με την Άστον σε μια άλλη έκθεση και ήταν τόσο πάρα πολύ δύσκολο να συλλέξει κανείς καν τα στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν αυτό έχει βελτιωθεί ή όχι. <clears throat> και ποιε είναι οι συστάσεις που θες να μας δώσεις, τις οποίες μπορούμε να υποστηρίξουμε όλες μας. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην ομιλητριά μας και θέλω να σας ζητήσω να είστε λίγο σύντομοι, γιατί έχουμε και άλλους εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα λάβουν το λόγο. Το υπόλοιπο τμήμα θα το προεδρεύσει η κυρία Σφέντσον Μπορώ να είμαι σύντομη, γιατί είναι απλές οι απαντήσεις. Η Γιούλεξ στο, Κοσο, στο Κοσφοπέδιο. <clears throat> έχω πάει διάφορες φορές εκεί, έχω συνεργαστεί με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Καταρχήν, η Ulex είχε τη δυνατότητα να έχει μία μονάδα για τα θέματα του φύλου. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήδη. Σαν άτομο και σαν εξάρτητο άτομο μπορώ να πω, ξέρω ότι υπήρξαν πολλά προβλήματα αλλά υπήρξε μεγάλη υποστήριξη σε υψηλό επίπεδο για αυτά που προσπαθούσε να κάνει η ομάδα για τα θέματα των φίλων. Αυτή ήταν η εντύπωση που σχήματισα εγώ. Επίση, υπήρξαν επαφέ με ομάδε γυναικών, επιτοπίου, επιτοπίους και μου δώσαν την εντύπωση ότι του εντυπωσίασε η λειτουργία αυτή τη ε, αποστολή Θεωρούν ότι χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη προσπάθεια σε ανθρώπινε σχέσει, σε δημόσιε σχέσει και μέσα σε αυτή την αποστολή και όχι. Αυτό που είπατε για την Βόρεια Ελλανδία, αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε περιλάβει στη μελέτη μας και αυτό φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και ζητώ συγγνώμη που δεν το έχουμε συμπεριλάβει. Το μεγάλο πρόβλημα τώρα με τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε πάντα όπου αυτό είναι απαραίτητο. Οπότε έχει πάντα κάνει στην εδώ επεκφυγής. Η πρόσβαση στα στοιχεία είναι καλύτερη, απαντώ στην κυρία Μπράντερ. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάστηκε να ρωτήσω και να ζητήσω πάρα πολλέ φορέ, ιδίω στην Κομισιόν, για να πάρω όλα αυτά τα στοιχεία για το προσωπικό. Δεν βρίσκονται αποθηκευμένα κάπου αυτά τα στοιχεία, δεν <clears throat> είναι ότι δεν θέλουν να μου τα δώσουν, αλλά δεν ξέρει κανείς πού βρίσκονται αυτά τα πράγματα. Το Συμβούλιο ήταν κάπως καλύτερο, αλλά όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν το την Ευρωπαϊκή Ένωση στο EAS να λειτουργήσει καλύτερα. Ποιο είναι αρμόδιο για αυτά, λέει κυρία Μπράντερ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μπαχαλώδη κατάσταση. Ο καθένα δεν ξέρει. Λέει για κάποιον άλλο. Βρίσκονται σε διάφορα email και σε διάφορα ε, έγγραφα, γιατί θέλω να θέσω ένα ερώτημα στη συνέχεια για το EAS. Ευχαριστώ πολύ. Η Εύα Μπρίτη να συνεχίσει την ε, προεδρία της συνεδρίασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ και την προσκεκλημένη μας. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε από την κυρία Γκία. Είδαμε τι στοιχεία υπάρχουν. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, θα ήθελα να καλωσορίσω κι άλλους εμπειρογνώμονες. Να υπενθυμίσω όμως ταυτόχρονα ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Έχετε όλοι 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Επομένως σας παρακαλώ πάρα πολύ μην ξεπεράσετε το χρόνο αυτό. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την κυρία Ντάγμαρ Σούμάχερ, που είναι η νέα διευθύντρια του Ινδιφέμ στις ε, Βρυξέλλες είναι το UN Women, του, ένα παρακλάδι αν θέλετε των Ηνωμένων Εθνών και θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Εύα, λέει η κυρία Σουμάχερ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Χάιντι που με κάλεσε. Είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την, ε, για την προηγούμενη παρουσίαση. Όμως ε, εγώ να σας μιλήσω τι έγινε τον Οκτώβρη είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αμήνας για τον 1325 και τα όσα έγιναν στη Νέα Υόρκη. Ε, έχουμε πάρα πολλά ε, κείμενα αν θέλετε, έχουμε στο χαρτί, στα χαρτιά έχουν γίνει πολλά πράγματα το πρόβλημα είναι τι έχει εφαρμοστεί. Εκεί χωλαίνει η υπόθεση. Λοιπόν, η πρώτη, ε, το πρώτο συμβάν για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω είναι για την συνάντηση που έγινε στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 13 ε, Οκτωβρίου και ε, εκεί αναφέρθηκε η παρουσία των γυναικών στις προσπάθειες ειρήνευσης και η συμμετοχή των γυναικών και στις ε, κυβερνητικές δομές. Ο Γενικός Γραμματέας επίσης ε, θεωρεί ότι είναι ευπρόσδεκτος στόχος ε, η η αύξηση της παρουσίας των γυναικών σε προσπάθειες ειρήνευσης από το 5% που είναι τώρα να φτάσει στο 15% και θα υπάρχει και η αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ε, όλα αυτά τα σημεία ε, αφορούν το τι μπορεί να κάνει ο ΟΗΕ και το σύστημα του ΟΗΕ. Αυτό ήταν ένα σημαντικό γεγονός η συνάντηση δηλαδή στις 13 Οκτωβρίου. Η δεύτερη σημαντική συνάντηση ήταν η ανοιχτή μέρα στις 21 ε, Οκτωβρίου του 2001, η ανοιχτή μέρα στη, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ε, εκεί συμμετείχαν διάφορες ε, οργανώσεις ε, γυναικών. Το ακούσαμε αυτό πόσο σημαντικό είναι από την κυρία Λούνατσικ προηγουμένως. Διάφορες γυναικείες οργανώσεις συμμετείχαν. Ήταν ένα κομμάτι των 27 ανοιχτών ημερίδων που είχαν οργανωθεί σε όλο τον πλανήτη μας από το Σουδάν, από το Νεπάλ και από το Μπουρούντι ήρθαν τρεις γυναίκες ε, ηγέτιδες, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και διάφοροι άλλοι υψηλοί αξιωματούχοι του ΟΗΕ. Η αίθουσα ήταν γεμάτη από πρέσβεις από το, το Συμβούλιο Ασφαλείας, από την εκπρόσωπη των, ε, της κοινωνίας, και είναι πάρα πολύ, ήταν πολύ σημαντική η συνάντηση αυτή και θα θέλαμε να θεσμοθετηθούν τέτοιου είδου εκδηλώσει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συμμετοχή των γυναικών, ε, η ενδυνάμωση του ρόλου, ε, του ρόλου τους στα θέματα διακυβέρνησης και επίλυσης των διενέξεων, ε, ο ρόλος των γυναικών κατά τη διάρκεια και μετά των, της ε, χρηματοδότηση, πόροι ε, για την ε, υποστήριξη των γυναικών στις διαδικασίες ανάκαμψης, αν θέλετε. Και το τελευταίο γεγονός, η τελευταία εκδήλωση για την οποία θα ήθελα να σας μιλήσω, αφορά την συνάντηση στις 26 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας αναγνώρισε ότι πολλά περισσότερα πράγματα θα πρέπει να γίνουν για να εφαρμοστεί ο 1325. Ε, αναγνωρίζει ότι διάφοροι δείκτες ε, θα πρέπει να δημιουργηθούν έτσι ώστε να παρακολουθούμε την θέση των γυναικών και στα θέματα ασφάλειας και οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και στην έκθεση του, Γενικού Γραμματέα προς το Συμβούλιο θα πρέπει να οργανωθεί καλύτερη δουλειά για τον 1325. Χρειάζεται στρατηγικό σχεδιασμό με βάση το 1325 και θα πρέπει τα επόμενα χρόνια, το επόμενο, το επόμενο έτος αυτό να γίνει. Και ε, θα ήθελα να μιλήσω λίγο παραπάνω για το τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση. Η συνάντηση αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας η κράτησε περισσότερο από ότι οι προηγούμενες συναντήσεις στην ιστορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, πάνω από 12 ώρες και συμμετείχε ένας ε, μεγάλος αριθμός ομιλητών, 91 συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα, της Μισελ Μπασλέ, που, στην οποία αναφερθήκαμε σήμερα, και παρουσιάστηκε η έκθεση του Γενικού Γραμματέα και αναγνώρισε την, ε, τα όσα έχουν κάνει τα κράτη-μέλη για τον 13-25. Μετά είχαμε ε, τον απληρωτή Γενικό Γραμματέα για τα θέματα διατήρησης της ε, ειρήνης. Συμμετείχαν ε, οι οικονομικές, εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών, του ΝΑΤΟ και πολλές χώρες συμμετείχαν με τους Υπουργούς Εξωτερικών συμπεριλαμβανομένης και της Χίλερου Κλίντον. Έγινε επίσης ε, και μια προεδρική δήλωση όπου χαιρετιζόταν ε, η δημιουργία του ΟΗΕ για τις γυναίκες ε, και ο διορισμός της κυρίας Μπασλέ και ενθαρρύνονται οι γυναίκες να, εργαστούν στα θέματα ασφάλειας και να παίξουν έναν ε, σημαντικό ρόλο στις ε, προσπάθειες ε, επίλυσης των διενέξεων. Και αναφέρεται επίσης και η ανάπτυξη, η ανάγκη δημιουργίας και ανάπτυξης αυτών των δικτών για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε κατάλληλα τον 13-25 λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαιτερότητα των κρατών μελών. Επίσης ε, ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τους και να εφαρμόσουν τους δείκτες που αναφέρονται στο παράρτημα. Αυτό αφορά και τα κράτη, το, της, ε, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε 26 δείκτες αυτή τη στιγμή, ε, εκ των οποίων οι 8 μπορούν να παρακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης από πλευράς κρατών μελών. Κάποιοι άλλοι δείκτες θα πρέπει να εφαρμόζονται από το σύστημα, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, από το UN Women. Αλλά εμείς θέλουμε δείκτες οι οποίοι, οι οποίοι να εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό, αυτή η προεδρική δήλωση δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στην ε, ελπίδα ότι το Συμβούλιο θα βελτιώσει το σύστημα όσον αφορά την, ε, το, την, την, την, ευθύνη και το σε ποιον υπόλογο ε, το Συμβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχει συνεπής εφαρμογή του 1325 και να εφαρμοστούν οι διαδικασίες παρακολούθησης. I would now like to look again. I mean, this this is maybe a bit uh, the reflection on the on the three events in October. Αυτά όσον αφορά τις τρεις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα τον Οκτώβρη. Τώρα, να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Τι χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι σαφές. Ε, από τη σημερινή μας συζήτηση. Χρειαζόμαστε πολιτική θέληση, ε, θέλουμε στοιχεία και δεδομένα ε, και χρειαζόμαστε πόρους και χρειαζόμαστε και ένα σύστημα που θα μας επιτρέπει να, να υπάρχει ένας καταμερισμός ευθυνών. Τώρα όσον αφορά τις άλλες δραστηριότητες και εδώ έχουμε πολλά να πούμε. Μιλήσαμε για τα εθνικά προγράμματα δράσης. Δεν έχουμε 27 εθνικά, ε, ε, εθνικά προγράμματα. Καιρός είναι να δημιουργηθούν και τα 27 ε, εθνικά σχέδια δράσης. Δεύτερον, Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας, κάτι το οποίο προβλέπεται, αυτό θα είναι ιδιαίτερα ευπρόζεκτο. Ένας πολύ συγκεκριμένος, ε, μια πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση των δικτών. Επίσης, εάν δείτε τι έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη όπου ε, ήταν η μέρα δέσμευσης θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε αυτό το παράδειγμα και στην Ευρώπη. Δηλαδή να υπάρχει μια ημέρα δέσμευση για κάποια συγκεκριμένα θέματα, να δούμε τι έχουμε πετύχει για το συγκεκριμένο τομέα και τι άλλο μπορούμε να πετύχουμε. Επίσης, ε, θα μπορούσαμε να δικτυωθούμε, θα μπορούσαμε να, να, να, συνεργαστούμε περισσότερο με τις ε, τοπικές οργανώσεις ε, και τους τοπικούς φορείς που ασχολούνται με τη θέση των γυναικών σε περιόδους και σε περιοχές ε, ε Εκεί νομίζω ότι εάν υπάρχει ε, μια πιο αποτελεσματική συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ε, τα πράγματα θα είναι καλύτερα και θα εξοικονομήσουμε και πόρους. Αλλά νομίζω ότι εξύντρισε το, χώρο, το χρόνο μου. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Ακούσαμε λοιπόν και καταλάβαμε μάλλον τους οκτώ σημαντικούς δείκτες για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Κατερίνα Λέιλονεν που εργάζεται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κυρία Λέινονεν είναι υπεύθυνη στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της 1325. Κυρία Λέινον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω κάποια λόγια για την εφαρμογή του 1325 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ καλό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση και ήταν τόσο δραστήριο και η κυρία Κία στη μελέτη της έδειξε ότι ήταν το πρώτο θεσμικό όργανο μετά την υιοθέτηση της 1325 που ξεκίνησε να προωθεί την εφαρμογή αυτού. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που είμαι εδώ σήμερα. Πολύ έγκαιρα γίνεται αυτή η συνεδρίαση. Πριν από 13 μέρες στη Νέα Υόρκη ε, έλαβε χώρα η ανοιχτή συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, κάτι που αναμενόταν ήταν αναμενόμενο γεγονός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ δραστήρια κατά την ε, περίοδο προετοιμασίας της συνόδου αυτής και πρόθεσε την υιοθέτηση των ε, δικτών, των γενικών δικτών από το ΟΗΕ που ετοιμάστηκαν με τη συνεργασία της UNIFEM και Τσοσάκη και έγιναν και διάφορες διπλωματικές επαφές και διαβήματα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για αυτόν τον σκοπό. Η δέκατη επέτειος συζητήθηκε επανειλημμένα σε διάφορες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου που διατύπωσε συγκεκριμένη θέση Ευρωπαϊκής Γιατί το λέω αυτό. Διότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς εφαρμόζουμε την ολιστική προσέγγιση κάνοντας χειρονομίες προς τα έξω αν θέλετε πλησιάζοντας τους έξω φορείς και πλησιάζοντας και τον ΟΗΕ. Όμως τώρα Αφού πέρασε αυτή η εκδήλωση, ελπίζω να προχωρήσουμε πιο πέρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και η Αυστρία σε αυτήν την συζήτηση ζητούσε ένθερμα έναν μηχανισμό γενικό για ενημέρωση υποβολή αναφορών και να υπάρχει ωστός μηχανισμός στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οπότε είναι πολύ ενεργή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται να αναφερθώ εκτενώς στην πολιτική μας, διότι η κυρία Χάουταλα και η κυρία Κία αναφέρθηκαν σε αυτό αλλά το 2008 ήταν η μεγάλη έκρηξη αν θέλετε εδώ και δύο χρόνια με πολύ ενδιαφέρον πολιτικό άνοιγμα και πρόθυμη γαλλική προεδρία που ήθελε να προωθήσει το θέμα αυτό και θεωρούσα πάντα σαν βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως την ειρήνη και την ασφάλεια και θεωρούσα ότι είναι σωστή η ολιστική γενική προσέγγιση και το, θα θα έπρεπε να δούμε πώς εφαρμόζεται 1325-1820 στην ΚΕΠΑ και οι κατευθυντήριε γραμμέ Ευρωπαϊκή Ενώσεω για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη βία κατά των γυναικών σημαντικοί πυλώνε. Δεν θα έπρεπε να μιλάμε πλέον για πυλώνε, διότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που είναι μετά τη Λισαβόνα, μετά τι Σύραξη. Μεταλισαβωνικό περιβάλλον. Λοιπόν, α μπούμε σε κάποια βασικά σημεία. Πάντα είναι καλό να αναφέρεται κανείς σε επιτεύγματα. Αν έχω χρόνο θα αναφερθώ και σε κενά. Ήδη τα ανέφερε η Κυριακία. Έχουμε 13 αποστολές, έχουμε συμβούλους σε όλες τις αποστολές για την ισότητα των φίλων και σε κάποιες αποστολές όπως UPOL Congo ή ULEX Κωσυφοπέδιο έχουμε πολλούς εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέματα που αφορούν την ισότητα των φίλων. Ενδιαφέρον παράδειγμα. Ήμουν στο UPOL Congo στην Κόμα το 2010 και εκεί είχαμε ένα αστυνομικό που ήταν επικεφαλής αντιπροσωπείας τρία μέλη της κινητής ομάδας σε σεξουαλική βία και έναν εμπειρογνώμη με τα ανθρώπινα δικαιώματα ισότητα των φίλων Και όλοι εργαζόταν για την USEC Κονγκό. Και τότε θεωρήσαμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θέματα των φύλων ήταν το βασικό ποσοστό ε, των προσπαθειών που καταβαλόταν στο Βορειοκιβού. Ετοιμάζουμε τα ε, ε, μια έκθεση σχετικά με τα μαθήματα που αντλήσαμε όσον αφορά τι αποστολέ και τα ανθρώπινα δικαιώματα ισότητα των φύλων είναι το πρώτο θέμα θα καλυφθεί. Ετοιμάσαμε πρώτο σχέδιο εκθέσεως. Και περνάει σε διάφορε ομάδε εργασία. Πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Διότι στι διάφορε ομάδε εργασία συμμετέχουν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι συζητήσει. Και σκεφτόμαστε τι δράσεις απαιτούνται και τι προτεραιότητα θα έχουν στο εγγύς μέλλον. Οπότε είναι πολύ επίκαιρη και η σημερινή μας συνεδρίαση για αυτόν τον σκοπό. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε επί του θέματος της κατάρτισης. Η Σουηδική Προεδρία πέρσι το πρόθεσε το θέμα. Τώρα θέλουμε να ετοιμάσουμε και διάφορα μοντέλα. Θα έχουμε διάφορα μοντέλα κατάρτισης για τα παιδικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα των φύλων στην διαχείριση των κρίσεων και ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα αυτά. Υπάρχει ιστοσελίδα για τις γυναίκες ειρήνη και ασφάλεια και ευκολία δυσκολία η ευκολία δυσκολία πρόσβαση στις πληροφορίες είναι κάτι που αναφέρθηκε εδώ. Ελπίζουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες. Έλεγχος. Οι εννέα δείκτες που ανέφερε η κυρία Κία ήταν η αρχική εκδοχή αυτών. Αρχές του έτους. Τον Ιούλιο υιοθετήσαμε 17 δείκτες προόδου όσον αφορά τη δική μας εφαρμογή του 1325. Σχετικά με την ΚΕΠΑ, διαχείριση κρίσεων και διαδικασίες ειρήνευσης. τι γίνεται και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των καταστάσεων που ακολουθούν συγκρούσεις και την πρόθεση της ειρήνης πώς κινούμεθα, προσμετρώντας και κατά πόσο το προσωπικό μας διαπράττει σεξουαλική εκμετάλλευση ή σεξουαλική βία. Θέλουμε αυτό να συζητηθεί ανοιχτά. Και ίσως δίνουμε ένα παράδειγμα να το κάνουμε αυτό. Τώρα εργαζόμαστε επί της εκθέσεως. Τις επόμενες εβδομάδες θα τελειώσει η έκθεση. Έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα τώρα σχετικά με το τι κάνουμε. Καλύψαμε και τους θεσμούς, αλλά και περίπου 20 κάτι μελη που μας απάντησαν. Άρα έχουμε ενδιαφέρουσα βάση δεδομένων. Κατανοούμε από τις παραληφθείς απαντήσεις ότι το 2009, αρχές 2010, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κάτι μέλη αυτής χρηματοδότησαν διάφορα προγράμματα σχέση με το 1325 σε 67 χώρες. Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ διατέθησαν. Θα δώσουμε πολλά παράδειγματα σχετικά στην έκθεση μας όπως η υποστήριξη που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σομαλία για τη δημιουργία προγράμματος για τις γυναίκες στη Σομαλία με τη συμμετοχή των διαφόρων φυλών. Αχ, περνάει ο χρόνος γρήγορα. Χαίρομαι που η UNIFEM είναι εδώ και ετοιμάζουμε σχέδιο υποστήριξης. Οι γυναίκες πέρα από τις συγκρούσεις και γεφυρώντας τη διάφορα ψηφίσματα του ΙΕ για την ε, ειρήνη και την ασφάλεια. Και ανοιχτέ ημερίδε αναφέρθηκαν επίση. Εμπνευστήκαμε από τον ΙΕ. Ζητήσαμε όλε τι αντιπροσωπείε μα σε έφταστε χώρε που έχουν περάσει σειράξει και σε αποστολέ και ΕΠΑ να ετοιμάσουν ανοιχτέ ημερίδε με τη συμμετοχή γυναικείων οργανώσεων. Εγώ ενθουσιάστηκα από τα αποτελέσματα. Συμμετείχα την περασμένη εβδομάδα μέσω του Skype σε μια συνεδρίαση σε μια μακρινή πόλη της Γεωργίας, όπου η αντιπροσωπεία μας εκεί, η αποστολή μας, είχε μαζέψει επιφανείς γυναίκες που ήταν σημαντικές στο επίπεδο το οικονομικό και το πολιτικό, για να συζητήσουν πώς τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά και στο Έρμπιλ στο Ιράκ θα γίνει άλλη συνεδρίαση αύριο με 150 συμμετέχοντες και αργότερα το μήνα αυτό στη Βαγδάτη. Μίλησα με την αντιπροσωπεία μας στη Βοσνία. Εκεί οργάνωσαν τέσσερις συναντήσεις σε όλη τη χώρα μαζί με τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Πολλά καλές ιδέες απέρευσαν από αυτό για τη συνεργασία επικεφαλής αντιπροσωπείας δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τη 16ημερη εκστρατεία που θα γίνει στη Βοσνία για την βία κατά των γυναικών. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα από αυτή την πρωτοβουλία που την αντιγράψαμε, μάλλον την αντιγράψανε μας τον ΙΕ, με την Αφρικανική Ένωση. Καλώ εταίρο η Αφρικανική Ένωση. Οργανώσαμε εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, παραδείγματο χάρη. Και τακτικά το θέμα της ειρήνης των γυναικών και της ασφαλείας συζητήσαμε στο διάλογο μας και διοργανώθηκε στην Αντίσα Μπέμπα για διήμερο εδώ και 15 μέρες. Στην Αντίσα Μπέμπα συνεδρίαση για μια ολόκληρη μέρα συζητούσαν το 13-25. Η κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης και της Αφρικής συμμετείχε εκεί. Υιοθετήσαμε πολλές συστάσεις και θα γίνει χαρτογράφηση του χρόνου, ε, χαρτογράφηση της εφαρμογής του 1925 στην Ευρώπη και την Αφρική. Και θα δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την κατάρτιση Αφρικανών ειρηνευτών και των διαφόρων ειρηνευτικών δυνάμεων. Τελείωσε ο χρόνος μου, δεν μπορώ να αναφερθώ στα κενά και στις συστάσεις θα αφορούσαν όμως την κατάρτιση, στελέχωση και πολύ σημαντικό ρόλο για τη νέα δομή που θα δημιουργηθεί. Και αναφορά στις θετικές εξελίξεις του διορισμού της, ε, προ... της Μάρσταν που είναι υπεύθυνη για το Σουδάν που πήγε ειδικά στην Αμπίσα Μπέμπα εδώ και 15 μέρες για να συναντηθεί με γυναίκες που ήρθαν από γειτονικέ χώρες του κέρατος της Αφρικής για να ακούσει τι έχουν να πούν. εντυπωσιακό Καλή κίνηση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λένονεν. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και κατέδειξαν σαφώς τι γίνεται και τι έχει γίνει στο παρελθόν και επομένως με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα αυτά τα οποία είπατε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λένα Αγ, που είναι Γενικός Γραμματέας μιας μη κυβερνητική σουηδικής οργάνωσης που έχει σαν ε, τίτλο «Κβίνα τιλ κβίνα, γυναίκες για τις γυναίκες». Είναι μια οργάνωση η οποία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα Βαλκάνια, με τον Κάυκασο, με την ε, Πρόσω Ανατολή και Πρόκειται για υποστήριξη οργανώσεων γυναικών που αγωνίζονται για να ενισχύσουν τις δυνατότητες της ε, γυναίκης. Δεν ακούγεται δυστυχώς η πρόεδρος γιατί έχει κλείσει το μικροφωνό της. Η κυρία Ακ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων και επίση και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πρόσκληση που μου απευθύνεται. Ελπίζω την επόμενη φορά θα ενδιαφερθεί και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εκπροσωπώ την, ε, το Ίδρυμα Κρίνα Τιλ Κρίνα, υποστηρίζουμε τις γυναίκες, τις οργανώσεις γυναικών επιτόπου σε περιοχές βίαιων συγκρούσεων για την βελτίωση των ε, δραστηριοτήτων τους. Ε, εμείς έχουμε τώρα και μια πλατφόρμα 28 οργανώσεων από 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΚΛΟ, η οποία εργάζεται και στον τομέα της οικοδόμησης ειρήνης και πιστεύω ότι έχετε και την ε, σειρά των προτάσεων μας για την εφαρμογή της 1325 τα 10 μας σημεία. Πριν από δύο εβδομάδες, <clears throat> μαζί με άλλες γυναίκες που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών από όλα τα τμήματα του κόσμου, ήμασταν παρόντες στην ανοιχτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το 1325, 13 χρόνια μετά από την αρχική έγκριση του ψηφίσματος αυτού, ήταν εντυπωσιακό ο κατάλογος των ομιλητών, όπω είπε και η Ντάκμαρ προηγουμένω. Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς <clears throat> ότι επειδή έχουμε ένα τόσο εντυπωσιακό κατάλογο αγοριτών, υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση για να ενισχυθεί ο ρόλο των γυναικών σε συνθήκε σύγκρουσης. Αλλά στην πράξη η επιτόπια κατάσταση παρά τη ρητορική δεν είναι πολύ καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Βλέπουμε σαν παράδειγμα, να έχουν περιθωρικοποιηθεί πλήρω οι γυναίκε στο Αφγανιστάν στι συζητήσει που γίνονται για την ειρήνευση εκεί πέρα. Αλλά η κατάσταση των γυναικών έχει γίνει πολύ χειρότερη μετά από τη στρατιωτική παρουσία σε αυτήν την χώρα. Η διάφθοση τώρα τη ομιλία μου είναι η εξή. Καταρχήν θέλω να ε, παρουσιάσω ορισμένε από τι εμπειρίε του δικτύου Κβίνα Τιλ Κβίνα. Θέλω επίση να σα αναφέρω ορισμένε ανεξάρτητε εκθέσει τη κοινωνία των πολιτών για το σε ποιο βαθμό τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη-μέλη έχουν συμπεριλάβει τις γυναίκες στην οικοδόμηση της ειρήνης <clears throat> και θα έχουμε συγκεκριμένες συστάσεις για τα κράτη-μέλη και για τον ΟΗΕ για να μπορούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο να προωθήσουν μόνιμη ειρήνη. Οι συστάσεις μας είναι απλές και ζητούν και την αντίστοιχη χρηματοδότηση. το ψήφισμα των γυναικών, όπως αναφέρεται ορισμένες φορές, το ψήφισμα 1325 των, του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει να κάνει με την ειρήνη και την ασφάλεια και αφορά τη συμμετοχή των γυναικών ως προαπαιτούμενο για την επέταξη της ειρήνης. Και επομένως συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία ειρήνευσης, τη συμπέριληψη της δικής τους οπτικής γωνίας μέσα στα πλαίσια της ουσίας των διαπραγματεύσεων. Εμείς θέλουμε να έχουμε πραγματικά μόνιμη ειρήνη. Είναι θέμα ασφάλειας και ειρήνης. Και πρέπει να υπάρχει σεβασμός των γυναικών και των δικαιωμάτων τους και αυτό αποτελεί αναγνώριση του γεγονότος ότι το ένα του πληθυσμού το οποίο υφίσταται βία ή διακρίσεις όσο είναι θύμα των συγκρούσεων δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη για κανένα και οι προκλήσεις και οι βιαιότητες κατά των γυναικών μπορεί να είναι αιτίε καταστροφής της ειρήνης και της ασφάλειας. Δέκα χρόνια μετά από την έγκριση του 1325 όμως φαίνεται ότι κανείς δεν ενσωματώνει μέσα στην πολιτική ασφαλείας του τις <clears throat> συστάσεις του 1325. Δεν έχουν μεταφερθεί στην πραγματικότητα. Γιατί, γιατί οι λήπτες αποφάσουν δεν ξέρουν πώς να εφαρμόσουν το 1325 ή ίσως γιατί ο χώρος αυτός κυριαρχείται από μια πολιτική ελίτ που είναι κατά πλειοψηφία ανδρική, που δεν κατανοούν τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών, τη σημασία της κατάστασης των γυναικών και το ρόλο που παίζουν οι γυναίκες σε όλα τα στάδια και τις φάσεις των ενόπλων συγκρούσεων. Επειδή οι γυναίκες περιθωρικοποιούνται από τις ιεραρχίες της εξουσίας σε μεγάλα μέρη του κόσμου, πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους για να έχουμε πολιτική επιρροή. Οι γυναίκε είναι πολύ καλέ στην οργάνωση, πολύ καλά κατανοούν τι ανάγκε των κοινοτήτων του και προτείνουν λύσει για τα προβλήματα αυτά και κατά τη διάρκεια και μετά από τι βίε συγκρούσει με έναν τρόπο που είναι πραγματιστικό. Όχι γιατί οι γυναίκε είναι πιο ειρηνικέ από του άντρε ή καλύτερε από του άντρε, αλλά γιατί οι επικρατούντε ρόλοι και η κατανομή των ρόλων για τα δύο φύλλα δίνουν στι γυναίκε τον προεξάρχοντα ρόλο για την οικογένεια και τα παιδιά. Μπορεί να νομίζει κανείς ότι αυτά είναι περισσότερο ανθρωπιστική και κοινωνική εργασία και όχι συμφιλίωση και ειρήνευση. Αλλά εμείς έχουμε την εμπειρία ότι με αυτές τις δράσεις οι οποίες γίνονται μπορούν αυτές οι δράσεις να οδηγήσουν σε διπλωματία μεταξύ απλών ατόμων. Παρά τις τραγικές τους λοιπόν απώλειες, οι γυναίκες σε εμπόλεμες καταστάσεις προσπαθούν να προωθήσουν το διάλογο και συνεργάζονται ακόμα και με τους πρώην εχθρούς τους στο Νότιο Κάφκας, όπου υπάρχουν πολλές λεγόμενες παγωμένες σειράξεις, οι γυναίκες είναι πάρα πολύ ενεργές στη διαδικασία ειρήνης και ε, συμφιλίωσης. Στην Αρμενία, παραδείγματος χάρη με τις γυναίκες Αζερί στον Αγκόνο Καραμπάχ και επίσης σε άλλες περιοχές του Καυκάσου μεταξύ Ρώσων και Γεωργιανών. Δυστυχώς, ε, πάρα πολλοί βλέπουν τις γυναίκες μονάχα υπό μία ιδιότητα ως θύματα. Είναι θύματα στις συγκρούσεις αυτές, αλλά το να βλέπουμε τις γυναίκες μονάχα σαν θύματα εμποδίζει να καταλάβουμε το ρόλο που μπορούν να έχουν οι γυναίκες και οι οργανώσεις τους για να παίξουν κάποιο ρόλο για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης. Και αυτό του βοηθάει πάρα πολύ τα πατριαρχικά συστήματα και τους αυτο, αυταρχικούς ηγέτες. Πολύ σπάνια οι γυναίκες φαίνονται ως οικοδομητές ειρήνες και υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γυναικών και ανδρών. Να σας φέρω τώρα ορισμένα πορίσματα της ανεξάρτητης έρευνας για την εφαρμογή του 1325. Τα έχουμε συζητήσει αυτά εδώ πέρα. Όλα τα πορίσματα δυστυχώς κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή ότι οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί δεν ε, τηρούν αυτά που υπόσχονται και δεν πραγματοποιούν αυτά που διδάσκουν. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτού το οποίο αναφέρει το 1925 και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα διπλωματικά κυκλώματα και τα προγράμματα για την οικοδόμηση ειρήνης. Τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγματι είναι καλά και θετικά, αλλά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται στην πράξη. Οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Αφρική και τη Μέση Ανατολή δεν έχουν λάβει υπόψη την συμμετοχή των γυναικών και εδώ βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε η Κέιτι Λέινονεν ότι τα πράγματα βελτιώνονται και εμείς έχουμε μια θετική αντιμετώπιση γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε οποιοδήποτε δυνατό τρόπο να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Περαιτέρω, κάποιο μέλος της Επιτροπής Ανέφερε πρέπει να αυξηθεί ο αριθμό των γυναικών που εργάζονται στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, η πρόοδο είναι πάρα πολύ βραδία. Θα ήθελα επίση ω ακτιβίστρια τη κοινωνία των πολιτών να υπογραμμίσω τον κέριο ρόλο που έχει να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα μπορούσε και ο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να προωθεί στο Κοινοβούλιο και τον έλεγχο της, της Κομισιόν και του Συμβουλίου όπως έχει πράξει στο παρελθόν. δεν <clears throat> μπορώ να σα υπενθυμίσω και δεν χρειάζεται να, το, να το υπενθυμίσει αυτό ότι μέσα στα πλαίσια της συζήτησης ε, για τις δημοσιονομικές προοπτικές μετά από το 2013 υπάρχει ανάγκη να δώσουμε προτεραιότητα στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται σε θέματα του φύλου και στις οποίες περιλαμβάνονται και ομάδες ε, γυναικών. και φυσικά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να διαδραματίσουν ένα κομβικό ρόλο και αναφέρθηκε προηγουμένως ότι τα περισσότερα σχέδια δράσης που περιλαμβάνουν τις γυναίκες για την ειρήνευση προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει όμως να τηρούν κοινά πρότυπα για να είναι αποτελεσματικά και στο έγγραφό μας για τα 10 σημεία που έχετε μπροστά σας αναφέρονται περισσότερα. Έχουμε τώρα στις τρεις συστάσεις για την προώθηση του ρόλου των γυναικών επί Πρώτον, να αναγνωριστεί σε πολιτικό επίπεδο αυτή η προσπάθεια. Οι γυναίκες ακτιβίτες πολλές φορές αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικέ απειλέ για την ασφαλεία του, αλλά δεν την χάνουν προστασίε. Ο αγώνα για την ειρήνη δεν είναι για αυτού οι οποίοι είναι ψοφοδέοι. Πολλέ φορέ υπάρχει μια τάση να χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές και να διαβάλλονται οι οργανώσεις των γυναικών. Είναι απαραίτητη η διεθνής αναγνώριση του έργου τους που θα μπορέσει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αξιοπιστία και προστασία. Θέλω να υπογραμμίσω ότι όλοι σας μέσα σε αυτή την αίθουσα έντιμοι βουλευτές και άλλοι πολιτικοί ηγέτες κάθε φορά που γίνεται σε μια περιοχή σύγκρουσης. <clears throat> Σας παρακαλώ να συναντήσετε με τις ομάδες των γυναικών, να μιλάτε μαζί τους, να παίρνετε πληροφορίες από αυτές. Θα βοηθήσετε πάρα πολύ να αυξηθεί το στάτους αυτό το όργανο. Στο δεύτερο, οι γυναίκε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε διαδικασίες ειρήνευσης και διαπραγματεύσει αυτή τη κατεύθυνση. 6% των διαπραγματευτών και 2% των μεσολαβητών μονάχα υπήρξαν γυναίκες τα τελευταία δέκα χρόνια διπλωματικών προσπαθειών για την ειρήνη. Ήρθε πια <clears throat> ο χρόνος να επιβάλλουμε πιστώσεις. Κάποιοι δεν συμφωνούν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε. Οι εμπειρίες των γυναικών χρειάζονται στις τάπεζες των διαπραγματεύσεων. Γιατί ο πόλεμος δεν τελειώνει με την τελευταία σφαίρα για τις γυναίκες. Και υπάρχει τώρα ένα παράθυρο ευκαιρίας μέσα εισαγωγικά σε κάθε συμφωνία ειρήνης να αλλάξουν οι ρόλοι των φίλων και να μην είναι μονοκόμματοι. Θέλω να κλείσω <clears throat> με την τρίτη μας, την τρίτη μου σύσταση και αυτή είναι φυσικά η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι σημαντική για την ανάπτυξη ικανότητος, για δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες και πολλές φορές οι γυναίκες που αγωνίζονται για την ειρήνη δεν καταφέρουν να έχουν χρηματοδότηση. Πολλά άλλα θα έλεγα, αλλά περιορίζομαι να πω ότι χρειάζεται μια ηγετικότητα και είναι καιρός να διοριστεί ειδικό εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων για τις γυναίκες και το ρόλο τους στις ένοπλες συγκρούσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν <clears throat> να γίνει κατανοητό ότι το 1325 δεν είναι για να γίνει ο πόλεμος ασφαλής για τις γυναίκες, αλλά για να έχουμε μια μόνιμη διαδικασία εξασφάλισης ειρήνης όλων τον κόσμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Αγ. Πράγματι, αυτό που είναι σημαντικό είναι το θέμα της χρηματοδότησης και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι μπορούμε να ακούσουμε ποιες είναι οι εμπειρίες του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό επιτρέπει τη βελτίωση των γνώσεών μας. Ευχαριστώ τους τρεις, τις τρεις προσκεκλημένες μας και ελπίζω να είστε έτοιμες να απαντήσετε και σε ερωτήσεις που θα θελήσουν να υποβάλουν οι βουλευτές. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Όποιος θα υποβάλει ερώτηση. Ε, η κυρία Λούνατζικ θέλει να ρωτήσει. Ναι, θέλω. Καταρχάς, από την Τίλα Κουίνα, η Φρανσέσκα Μπράντνερ και εγώ είμαστε συντονιστές Πρασίνους και είμαστε μέλη της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Είπατε ότι δεν είναι κανείς, είμαστε εμείς εδώ. Θέλω να είμαι λίγο προκλητική, όχι για τους παρισταμένους, αλλά έχω την εντύπωση καμιά φορά όταν γίνονται ψηφίσματα όπως για τις και την ειρήνη και την ασφάλεια, αισθάνομαι ότι έπρεπε να έχουν διαφορετική ονομασία όπως άντρες, γυναί... Ε, ε, άντρες ειρήνη και ασφάλεια διότι έτσι ώστε να ενδιαφερθούν περισσότεροι άντρε για το θέμα, όχι γιατί αφορά τι γυναίκε. Οι γυναίκε δεν είναι μόνο θύματα, είναι θύματα, αλλά είναι και αυτέ που οικοδομούν την ειρήνη. Ίσως να αλλάξουμε τη γωνία. Σαν φεμινίστρια Η μη προβολή των γυναικών. Η ασφάλεια και η άμυνα και εξωτερικές υποθέσεις κυριαρχούνται από τους άντρες. Ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά θέματα κυριαρχούνται από τις γυναίκες και χρειάζεται μια αλλαγή και εκεί. Τούτων λεχθέντων. Έχω ερώτηση προς την κυρία Λένανεν για την υπηρεσία εξωτερικής δράσεως. Η Φρανσίσκα Νερ και εγώ ενδιαφερόμαστε πολύ. Μπορείτε να μας πείτε ποια θα είναι η μελλοντική μορφή όσον αφορά τα θέματα ισότητας των φύλων. Στις επαφές μας με την κάθε Άστον, στις διαπραγματεύσεις, ζητούσαμε ότι η δομή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι κάτι βασικό και ισότητα των φίλων επίσης. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κατεύθυνση της δομής αυτής. Υπάρχει κάποια μορφή επικρατή σύγχυση. Σας ξέρω από το... Είσαι στο Συμβούλιο, εμείς Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το θέμα μας. Και το κοινοβούλιο πρέπει να σπρώξει για να γίνουν κάποια πράγματα. Και τα κράτη-μέλη επίσης πρέπει να προωθήσουν και η κοινωνία των πολιτών. Φαντάζομαι ότι και εσείς κάνετε τα ίδια. Πείτε μας κάτι πάνω σε αυτό. Από δική μου εμπειρία, εργάστηκα στην κοινωνία των πολιτών επί μακρόν πριν γίνω πολιτικός. Και είναι το θέμα των ποσοστώσεων που τίθεται. Αν δεν ζητήσουμε ποσοστώσεις, σχεδόν παντού, η ίσες διαπραγματεύσεις τουλάχιστον, δεν θα έχουμε την προβολή των γυναικών όπως θα έπρεπε. Δεν θα υπάρχει σωστή εκπροσώπηση των γυναικών, τόσο ώστε να υπάρξει πρόοδος. Σε πολλούς δεν αρέσει αυτό λένε ότι χρησιμοποιούνται γυναίκες ως άλοθη για τις ποσοστώσεις. Υπάρχουν και πολλοί άντρες όμως που είναι σε θέσεις επειδή είναι μόνο άντρες και όχι λόγω ικανοτήτων ή γιατί αντιπροσωπεύουν κάτι. Πολλοί στην ομάδα μου το υποστηρίζουν αυτό. Το συζητήσαμε και στο Κοινοβούλιο. Στις επόμενες εκλογές, στην επόμενη θητεία, ίσως και του χρόνου για κάποιες θέσεις που θα αλλάξουν, να ζητήσουμε περισσότερες γυναίκες, πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση στα Προεδρία των διαφόρων επιτροπών. Αυτά. Stort Ευχαριστώ πολύ κυρία Λούνατζεκ. Θα μπορούσαμε να πούμε, λέει η κυρία Σβένσον, ότι ένας από τους λόγους για τις οποίους ε, οι γυναίκες ε, αντιμετωπίζονται σαν θύματα δεν εξαρτάται δεν εξαρτώνται από την κατάσταση αυτή αυτή από την περίπτωση, αλλά γιατί τις βλέπουν τις γυναίκες μόνο και αποκλειστικά στο ρόλο του θύματος, χωρίς να εξετάζουν τις δυνατότητες που έχουν να συνεισφέρουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο σε ορισμένες περιστάσεις να αντιμετωπίζονται οι γυναίκες απλώς και μόνο σαν θύματα, χωρίς να βλέπουμε τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να προσφέρουν. Τώρα, όσον αφορά τις ε, ποσοστώσεις, η, η επίδραση και η παρουσία των γυναικών στην, ε, στην Επιτροπή μας, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και του χρόνου θα ξανασυζητήσουμε το θέμα Άρα ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζονται προφανώς περισσότερες γυναίκες στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες να δείξουν αλληλεγγύη μεταξύ τους. και να υποστηρίζουν ε, τις γυναίκες που αναλαμβάνουν ε, αρμοδιότητες. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε και εμείς σαν γυναίκες ε, τις γυναίκες που θα αναλάβουν κάποιες θέσεις, κάποια αξιώματα, κάποιες αρμοδιότητες. Θα ήθελα να σας τώρα το λόγο και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, διότι δεν είπα σωστά το όνομά σας. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μία ερώτηση να κάνω όμως, που ίσως είναι αυτονόητη. Αλλά υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ένα αντίστοιχο των εθνικών σχεδίων ε, για την εφαρμογή του 1325 και μήπως χρειαζόμαστε και ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του 1325. Ευχαριστώ, κύριε Κορνίλισεν. Συνήθως ε, μιλάει κάποιος ε, εξ κάθε ομάδας. Ε. Αλλά επειδή δεν είμαστε και πάρα πολλοί παρόντες και παρούσες, μπορούν και οι δύο εκπρόσωποι των πρασίνων να πάρουν το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομη και θα πρέπει να φύγω και σε ένα λεπτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλές παράλληλες συνεδριάσεις να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε η Λουρίκε. Θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα ε, σαν βουλευτές για να κάνουμε τη δουλειά μας να έχουμε περισσότερες ε, πληροφορίες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και που θα αφορούν ε, διάφορες χώρες οι περισσότεροι εξημών συμμετέχουν σε αντιπροσωπείες με διάφορα σημεία του πλανήτη μας και πιστεύω ότι πολλοί θα ήθελαν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, εάν και εφόσον βέβαια γνώριζαν και κάτι παραπάνω. Αλλά χρειαζόμαστε πληροφορίες συγκεκριμένες ε, που να αφορούν κάποια έκθεση ή κάποια επίσκεψη που θα έχει οργανώσει το Κοινοβούλιο στο εξωτερικό. Επίσης, θα θέλαμε να ακούσουμε και κάποιες προτάσεις σας για τροπολογίες που θα μπορούσαν να γίνουν ε, στις ε, εκθέσεις που συντάσσονται για κάποιες χώρες. Όσο πιο συγκεκριμένη είναι η πληροφορία, τόσο πιο εύκολο είναι για μας να την χρησιμοποιήσουμε στη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εγώ πραγματικά θα ήθελα ε, στην επόμενη έκθεση που θα κάνουμε για τα Βαλκάνια, όπου ε, αυτή τη στιγμή ε, ε, βρίσκονταν εξελίξει διαδικασίες ειρήνευσης. Και εγώ που ασχολούμαι με τα θέματα ισότητα των δύο φύλων εδώ και χρόνια και για τα δικαιώματα των γυναικών, δεν είχαν ερωτηθεί σε αυτές όλες τις διαδικασίες ειρήνευση ποιο είναι ο ρόλος των γυναικών, εκπροσωπούνται επαρκώ. Λοιπόν, θα ήθελα για όλα αυτά τα θέματα να ακούσω και την άποψη των εμπειρογνωμόνων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κορνίλσεν, λέει η κυρία Σβένσον. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο τώρα στους, στις τρεις ε, προσκεκλημένες μας. Ε, η κάθε μια από τις ε, τρεις θα έχει δύο λεπτά. Τον λόγο τον δίνω στην κυρία Σούμαχερ καταρχάς για να βγάλει τα συμπεράσματά της. Δεν νομίζω, Δεν νομίζω ότι έχω πολλά να προσθέσω. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που είπε η κυρία Κορνέλσεν και μπορούμε και εμείς να δώσουμε πληροφορίες από τη δική μας πλευρά. Και είναι ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ότι ακόμα και αν έχει δουλέψει κανείς σε αυτό το θέμα πολύ καιρό, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν τα σκέφτεται. Και πολλές φορές βλέπει κανείς αυτές τις συναντήσεις ότι το προφανές δεν είναι προφανές. Ε, πέραν τούτου, νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον αυτό που ελέγχθη για τα εθνικά σχέδια δράσης και αυτά μπορεί να είναι πράγματι ενδιαφέροντα να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράση, το οποίο θα είναι πιο πλήρε. Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που μπορώ να απαντήσω εγώ. Απλώ θα ευχαριστήσω για αυτήν την ιδέα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λέινον έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ αναφέρθηκα για, την, ε, για το περιφερειακό σχέδιο δράσης RAP της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια πλήρη αντιμετώπιση. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για το ποιος κάνει τι. Είναι χρήσιμο να έχουμε και ενδείκτες οι οποίοι καλύπτουν αυτά τα στοιχεία. Έχουμε ξεκινήσει όμως πολύ καλά και είχαμε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το 2008 να τα προωθήσουμε. Προς το παρόν λοιπόν αυτό είναι το σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές πληροφορίε για τη μελλοντική διάρθρωση που θα έχει η αντίστοιχη δομή των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν του οργανόγραμματος που είχε παρουσιάσει η κυρία Άστον, αυτό μου θύμισε πολύ το οργανόγραμμα της EU-LEX με γεωγραφικές διευθύνσεις και μετά μία διεύθυνση που ασχολείται μονάχα με πολυμερή θέματα και ένα από τα οποία ήταν το θέμα του των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το φύλλο. Δεν ξέρω όμως αν αυτή είναι η δομή η οποία θα εξακολουθήσει να ισχύει <clears throat> στο μέλλον. Αν έχει κανείς το, τη διάσταση του φύλλου μόνο σε μια δομή που είναι παράλληλη προς όλες τις άλλες, είναι πολύ δύσκολο να έχει το απαραίτητο ειδικό βάρος όλη αυτή η προβληματική με τις άλλες που ανταγωνίζεται τις άλλες δομές οι οποίες και αυτές εμπλέκονται στην ε, ιεραρχία. Οι δομές αυτές λοιπόν που τις γνωρίζει πολύ καλά η Κατερίνα Βάλεντου, τη συνάδελφος μου από το Συμβούλιο, όλες αυτές οι δομές έχουν μια κατευθείαν πρόσβαση στα υψηλότερα επίπεδα, κάτι το οποίο δεν είχαν οι άλλες διευθύνσεις. Και όταν είδαμε αυτή τη δομή Αναρωτηθήκαμε αν αυτό θα βελτιώσει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην ΚΕΠΑ. Ερωτηματικό. Ήθελα να πω κάτι περισσότερο, αλλά το ξέχασα. Οπότε θα σταματήσω εδώ. Α, το θυμήθηκα, το θυμήθηκα. Η δική μου εμπειρία <clears throat> από την Γενική Διεύθυνση ΡΕΛΕΞ για την ασφάλεια των γυναικών, μετά πήγα στο Συμβούλιο. Αυτό μου κατέδειξε πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ο ρόλος ε, του προσωπικού σημαντικός ρόλος του προσωπικού εκπροσώπου του Χαφιέ Σολάρα. Και εκεί είναι θέμα προσωπικότητας και χρειάζονται άτομα τα οποία να μπορούν να προωθήσουν αυτή την ατζέντα όπως έκανε τότε η εκπρόσωπος του Σολάνα γιατί είχαν το κύριο και την προσωπικότητα. Απλώς αυτό σας το αφήνω σε μία σκέψη. Ευχαριστώ κυρία Λέιτονεν και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Αγκά. Mm. Πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη αυτή και ίσως να δίνει και μια, ένα παράδειγμα, μια ιδέα στο Κοινοβούλιο τι μπορεί να επιτευχθεί όταν, ε, όσον αφορά την πρόθεση, όπου την είπατε εκπρόσωπο του 1925, όσον αφορά τι ποσοστώσει, γιατί είναι μακρά συζήτηση και ξέρω το Κοινοβούλιο ε, συνεχώς το εξετάζει. Οι ποσοστώσεις λειτουργούν, αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε και το είδαμε όσον αφορά την πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να το σκεφτείτε αυτό. Όσον αφορά τις πληροφορίες κατά χώρα, μπορούμε να δώσουμε τις πληροφορίες και ε, νομίζω ότι η αρμόδιος φορέας είναι πρόθυμος να δώσει τις πληροφορίες. Και έχουμε και το έγγραφό μας που αφορά, δείχνει τη θέση μας όσον αφορά διάφορα ζητήματα, όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα δράσης. Να πω ότι η σκανδιναβική. Και οργανώσεις κάναμε ταξινόμηση των σχεδίων δράσεως των σκανδιναβικών χωρών και η Φιλανδία ήταν η χώρα εκείνη που ίσως να σας ενδιαφέρει. Διότι ήρθε πρώτη. Όμως υπήρχαν προβλήματα γενικά που αφορούσαν την κατανομή των πόρων, συγκεκριμένους στόχους, προτεραιότητες, χρονοδιαγράμματα κλπ. Όταν μιλάμε για εθνικά σχέδια δράσης χρειάζονται κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές. Αλλά παρακαλούμε μην αφήνετε αυτά τα εθνικά σχέδια δράσης να εμποδίσουν τη δράση. Μπορούμε να σχεδιάζουμε αένα, αλλά πρέπει να κάνουμε και να κάνουμε περισσότερα από την άλλη. Τελικό μου σχόλιο, αυτό ήταν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Άγκ. Πριν να δώσω το λόγο στην κυρία Αουτάλα για να κλείσω. Νομίζω ότι η κυρία Σουμάχερ έχει κάποιο σχόλιο. Πολύ γρήγορα να προσθέσω κάτι που ανέφερε κάτι. Δεν θέλω να φύγω από εδώ πριν μπω. Ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έσπρωξε και προώθησε τον οδικό χάρτη προς έγκριση των δικτών ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ήταν πολύ σημαντικό τα κάτι μέλη υποστήριζαν αυτή τη θέση στις συζητήσεις που έγιναν στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύα Μπρίτ, αυτό δείχνει ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεργαστούν στενά με την γυναίκα ισότητα των φίλων και δικαιωμάτων της γυναίκας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι ακούσαμε πολλές καλές ε, συστάσεις, όπως η ιδέα ειδική εκπροσώπου. Πρόσφατα το συζήτησα το θέμα αυτό με τους επιτετραμένους ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως των διαφόρων Υπουργείων. Γιατί να μην έχουμε θεματικούς ειδικού εκπροσώπους, όπως έχουμε ειδικό εκπρόσωπο τη Ροζαλίν Μάστεν στο Σουδάν. ειδικοί εκπροσώπη για τα, ανθρώπινα, για τα γυναικεία δικαιώματα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα ήταν σημαντικό ίσως και για την συγκρότηση ειρήνης μπορεί να εξεταστεί σαν θέμα. Μπορούμε να συνδυάσουμε διάφορες στοιχεία στην προσπάθεια αυτή. Οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ενώσης θα μπορούσαν να ε, διαθέτουν κάποιους πόρους για τις προσπάθειες που καταβάλουν οι γυναίκες, για την ειρήνευση υποστηρίζονται πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό γίνεται σε άλλους τομείς με μικρές χορηγίες. Δεν πρέπει να υποτιμάμε το ρόλο των αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την πρόθεση της εικόνας των γυναικών. Προσωπικά μου αρέσουν οι ποσοστώσεις. Είδα ότι λειτουργούν στην πράξη. Έτσι οι ικανές γυναίκες μπορούν να προβάλλονται διότι το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά ε, δεν, τις, ε, δεν προωθούνται και δεν καταλαμβάνουν τις θέσεις και είναι καλές οι γι' αυτό. Ξεκινά αναθεώρηση τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είπα ότι εκπρόσωπο, μάλιστα ανέλαβε να τη δρομολογήσει αυτή. Ξεκίνησαν οι συζητήσει στο Κοινοβούλιο, ξεκινάνε μάλλον μεταξύ κρατών μέλων. Τα γυναικεία δικαιώματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην στρατηγική τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και γυναίκε και ειρήνη και συγκρούσει Χρειάζεται στενή συνεργασία με τις κοινωνίες των πολιτών. Και αναφέρεται ότι υπάρχουν διάφοροι αρμόδιοι για επαφές όσον αφορά τις ε, προσπάθειες για ειρήνευση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ, Εύα Μπρίτ. Ακούσαμε προτάσεις που μπορούν να μας φανούν χρήσιμες στην καθημερινή μας δουλειά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για αυτή την ενδιαφέρουσα απογευματινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ τους βουλευτές, τη γραμματεία. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. Ευχαριστώ όλους. Καλό σας βράδυ.